Välkomna. Uh, Καλώς ήρθατε. Έχουμε πάρα πολύ βαριά ημερήσια διάταξη και για σήμερα και για αύριο. Πριν την έγκρισή της θα ήθελα να κάνω τις εξής ανακοινώσεις για το σχέδιο ανάκτησης ε, της οικονομίας ε, της κυρίας Μογά, ανάκαμψης της οικονομίας. Θα κάνουμε αμέσως τώρα τη συζήτηση. Κανονικά ήταν να γίνει αύριο, αλλά θα γίνει σήμερα. Είναι γνωμοδότηση και πρέπει να τη δώσουμε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Γιατί αναμένεται αύριο η έγκρισή της, οπότε θα πρέπει να τη συζητήσουμε. Δεν, ε, η, κάρτα μου δεν λειτουργεί. Ε, θα ψηφίσω χωρίς ηλεκτρονική κάρτα. Ναι, Μα δεν μίλησα εγώ για τις κάρτες. Δεν το ξέραμε αυτό, οπότε θα ψηφίσουμε χωρίς κάρτες. Κανονική ψηφοφορία. Οπότε δεν πειράζει αν δεν έχουν κάποιοι τις κάρτες μαζί τους. Λοιπόν, μετά... Στο σημείο 20, παιδιά μεταναστών, ε, πρέπει να το συζητήσουμε κανονικά συνεδρίαση συντονιστών, αλλά Θα ασχοληθούμε με την ε, οδηγία για το χρόνο εργασίας ε, και είναι πολύ φορτωμένη η μερίσια διάταξη. θα το συζητήσουμε λοιπόν το θέμα σήμερα και θα ψηφίσουμε αύριο. Παρότι δεν το συζητήσαμε στους συντονιστές. Αυτές τις αλλαγές ε, θα κάνουμε μόνο. Μπορούμε να εγκρίνουμε τώρα το σχέδιο με εσείς διάταξη. Ευχαριστώ. Uh, what? Ja, vi, vi har protokollet ε, α, πρέπει να εγκρίνουμε και τα πρακτικά. Εγκρίνονται, ναι. Άλλες ανακοινώσεις τώρα. Υπάρχει web streaming σήμερα της συνεδρίασης. Επίσης, ένα μικρό κλιμάκιο μετέβη την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Εγώ και η κυρία Γέλεβα από το ΕΛΚ συγκεκριμένα και συναντηθήκαμε με υπαλλήλους του ΟΗΕ και συναντηθήκαμε και με την εκπροσώπου της Επιτροπής. Συζητήσαμε την μελλοντική συνεργασία της Επιτροπής μας εδώ στο Κοινοβούλιο με τον ΟΗΕ. Στο μέλλον θα ε, υποβληθεί και μια έκθεση από αυτή την αντιπροσωπεία από εμένα και από την κυρία Γέλεβα, δηλαδή για αυτή τη συνάντηση που κάναμε. Επίσης, ε, στην συνεδρία του Συμβουλίου, στο Λούχα Κόβιτσε, στις 22 και 23 Ιανουαρίου στη Τσεχία, ε, είχαμε στείλει μία αντιπροσωπεία και έχετε το αντίστοιχο σημείωμα. Και τέλος, Καλωσορίζω την κυρία Μαρλή Γεσόμπα, νέα συνεργάτηδα. Καλωσορίσατε. Ας τη χειροκροτήσουμε. All of you, Όλοι να χειροκροτήσουμε <laughs> Ευχαριστώ. Αυτέ ήταν οι ανακοινώσει μου. Πάμε στο πρώτο σημείο. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ανάκαμψη τη οικονομία. Η κυρία Μόχα είναι η συγγήτριά μα. Έχετε τον λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σα πω πριν αρχίζουμε να ψηφίζουμε ότι λάβαμε υπόψη μας συνολικά όλες τις παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη συμπιτροπή. Πιο συγκεκριμένα στην ε, βούληση όλων μας, ώστε τα ηλιμένα μέτρα να εγγυηθούν την απασχόληση των μισθωτών διότι είναι πολύ πιο εύκολο να κρατήσει κάποιος τον εργαζόμενο στην δουλειά όσο τον απασχολεί από ότι όσο να τον ξαναφέρει όταν δεν τον απασχολεί. Αυτό το σχέδιο ενάκαμψης επίσης θα πρέπει να χρησιμεύσει ούτως ώστε μέσα από σχέδια κατάρτισης να αναβαθμιστεί να αναβαθμιστούν και οι ικανότητες των εργαζομένων. Καταγράψαμε όλες τις παρατηρήσεις και μαζί με την κυρία Φερέρα και τους εκπροσώπους από τις άλλες αρμόδιες επιτροπές κάναμε συντονιστικές συνεδριάσεις συνεδριάσεις όπου ανταλλάξαμε απόψεις, συζητήσαμε, διότι καταφέραμε να οικοδομήσουμε, να φτιάξουμε όλοι μαζί συμβιβασμούς που θα ικανοποιούν όλα τα πολιτικά κόμματα. Να σας το πω όμως πολύ ειλικρινά ότι αυτές οι συνεδριάσεις, οι ε, συντονιστικές συνεδριάσεις μας επέτρεψαν μέσα από το διάλογο να σεβαστούμε τη, οι ιδέες των δε και η γνωμοδότηση όπως έχει σήμερα εύχομαι να σας ικανοποιεί τα μάλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Oh. Ευχαριστούμε, κύριε Μογά. Ο κύριος Σίλβα Πινέιντα η κυρία Κουζανικόβετς είναι στον κατάλογο των ε, ομιλητών. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ την, συγγητή, αλλά ε, δεν μπορώ παρά να τονίσω τους περιορισμούς ε, που υπάρχουν λόγω της οικονομικής κρίσης έχουμε, πρέπει να έχουμε επίγνωση της κρίσης ε, και με ακόμη και στο χώρο ε, της, ε, του ευρώ το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είναι ενιαίο. Υπάρχουν 27 διαφορετικά συστήματα. Δεν έχουμε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Έχουμε εθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν έχουμε μια μακροπρόθεσμη οικονομική πολιτική που μας επιτρέπει να ανταπεξέλθουμε παρκώς σε αυτή την κρίση. Οπότε τα προσεχή χρόνια η αυξανόμενη ανεργία ε, θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση της τιμής ε, του χρήματος και άρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν επενδύσεις ε, Λοχεύει αυτός ο κίνδυνος σε σχέση με την πίστη και αν συγκρίνουμε παραδείγματος χάρη ε, την ε, Γερμανία με την Ελλάδα βλέπουμε πόσο διαφορετικές ε, είναι οι επιστοληπτικές ικανότητες παραδείγματος χάρη και είναι πολύ ευπαθείς οι οικονομίες μας και θα πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες, να λάβουμε άλλου τύπου μέτρα, ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και θα πρέπει να βρούμε μία λύση η οποία παραδείγματο χάρη θα μπορούσε να βρεθεί στα χαμηλά επιτόκια επί σειρά ετών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιδόσεις των κρατών μελών και δύσκολα πλέον ε, τα κράτη-μέλη μπορούν να μαγειρεύουν τους λογαριασμούς όπως κάνανε στο παρελθόν. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εκδίδεται δημόσιο χρέος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με, την ίδια, με τον ίδιο βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας, αλλιώς ε, δεν προβηκείται να αντιμετωπιστεί ε, το πρόβλημα και της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας. Ξαναλέω ε, ότι η δημόσιο χρέος θα πρέπει πλέον να συνάπτεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να εξασφαλίσουμε τις επενδύσεις που χρειαζόμαστε. Αυτό σχετίζεται με αυτά που μας έλεγε η συγκήτρια, αλλά υπάρχει και με σε μια συμβαστική τροπολογία, δηλαδή για να καταπολεμήσουμε την οικονομική κρίση θα πρέπει οπωσδήποτε να διαρευνήσουμε αυτή τη λύση. Ευχαριστούμε η κυρία Κοζανικόβατζε. Κυρία Λέντρε Μάγδα στη συνέχεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου στην ε, εισηγήτρια γιατί πρόκειται για μια έκθεση που βασίστηκε σε πολύ καλό συντονισμό. Υπάρχει ένα πρόβλημα, όπως ξέρετε, τα κράτη-μέλη πρέπει να ξεπεράσουν τις ε, διαφορές ε, που έχουν και να συντονίσουν τα στρατηγικά μέτρα. Και όπου χρειάζεται αλληλεγγύη θα μπορέσουμε να βρούμε τη βάση για αυτή την αλληλεγγύη και αυτό αποδείχθηκε και στην διαδικασία σύνταξης αυτής της ε, έκθεσης που μπορέσαμε να συμβιβάσουμε τις ε, θέσεις μας. Οπωσδήποτε πάντα θα υπάρχουν διαφορές και καθώς ε, αρκετές χώρες ακόμα απέχουν πολύ από την Ευρωζώνη σημασία έχει να τονίσουμε πως αυτές οι διαφορές διαφορές ε, σε ευκαιρίες που έχουν οι χώρες πρέπει να μειωθούν. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι έτοιμο να υπερψηφίσει τις άλλαγες ε, ε, που έχουν προταθεί και για μία μόνο από αυτές έχουμε σοβαρές αμφιβολίες για το εάν είναι δυνατόν δηλαδή σε τρεις μέρες να δημιουργούνται εταιρείες στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε νομίζω λίγο περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αφού συγχαρώ και ευχαριστήσω την Ελιζαμπέτ Μογάν γιατί συνεργαστήκαμε εξαιρετικά υπό την καθοδήγησή της γύρω από αυτό το κείμενο, να σταθώ σε αυτό που είπε και η συνάδελφος Σίλβα Πενέδα. Είναι σαφές ότι αν δεν κάνουμε τίποτα στα πλαίσια της Ευρωζώνης θα αφήσουμε τις χώρες που βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση να δανειστούν με ψηλότερα επιτόκια. Αυτές οι χώρες λοιπόν οι οποίες θα έχουν περισσότερες δυσκολίες να προσθέσουν ακόμη δυσκολίες. Στην Ευρωζώνη λοιπόν θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να αποσύρει την ποσόστοσή του ο καθένας ή να μην την αποσύρει. Το δάνειο, η δανειοδότηση λοιπόν στο πλαίσιο της Ευρωζώνης είναι θεμελιώδης. Ευχαριστώ. Κανείς άλλος δεν έχει εγγραφεί στον κατάλογο. Κυρία Μογά, έχετε το λόγο πριν αρχίσει η ψηφοφορία. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, après vous avoir euh, tous écouté, de vous dire mes... Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ειλικρινέστατα. Να ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά τους εκπροσώπους ε, των πολιτικών κομμάτων που συνεργάστηκαν ώστε να καταλήξουμε επικοδομητικά σε σοβαρές προτάσεις σε αυτή τη γνωμοδότηση. Σε αυτό τώρα που είπαν οι συνάδελφοι Σίλβα Πενέδα και Λεϊντέ αυτή η πρόταση για ένα μεγάλο δάνειο στην Ευρωζώνη ούτω ώστε να μην δημιουργηθούν ανισότητες μεταξύ των χωρών. Εμείς σε αυτήν την πρόταση προσέξαμε να μην ξεπεράσουμε τις αρμοδιότητες μας ως Επιτροπή Επασχόλησης... Και όλη η εργασία που κάναμε σέβεται τις αρμοδιότητες μας σε αυτήν την Επιτροπή. Πάντως πρέπει να σας πω ότι ήμουνα πάρα πάρα πολύ προσεκτική ε, για στη συνεργασία μου με τους άλλους, ούτως ώστε να προσεγγίσουμε την συνένεση και να έχουμε μια θετική ψηφοφορία. Ευχαριστούμε. Πάμε στην ε, ψηφοφορία τώρα. Στίβεν και Φίλιπ, συντονιστές. <laughs> με Συμβαστική α υπέρ. Κατά. Μικρή διαφορά. Ξανά θα ψηφίσουμε γιατί δεν ξέρω από πλευρά σοσιαλιστών. Εντάξει, δεν ε, ξέραμε ότι θα γίνει ψηφοφορία σήμερα, γι' αυτό σας είπα θα ψηφίσουμε χωρίς κάρτες. Ξαναψηφίζουμε για τη συμβαστική Α, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Πολύ μικρή διαφορά, θα γίνει καταμέτρηση. Υπέρ πάλι για την συμβαστική Α. Κατά. Αποχές. Πενήντα υπέρ, 21 κατά, καμία αποχή. Ε, τροπολογία 1 τώρα, ε, της κυρίας Τόγια, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική Β. Σε δύο τμήματα παρακαλώ. Συμβαστική Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μου λένε ότι πρέπει να ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα μόνο της δεύτερης τροπολογίας, μόνο το πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική συν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. πίπτη η 3. Ψηφίζουμε την 4 τώρα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 8 αποσύρθηκε 9 σε τρία τμήματα πρώτο τμήμα calls for μέχρι το employment initiative υπέρ παρακαλώ για το πρώτο τμήμα κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα από το on the one hand μέχρι το three days. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά πρέπει να γίνει καταμέτρηση. Για το δεύτερο τμήμα ψηφίστε πάλι παρακαλώ υπέρ. Αποχέ. Ε, αποχές. Δεκαεννιά προς 17, καμία αποχή, οπότε εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα τώρα, and that the formalities μέχρι το businesses. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 12 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 καταπίπτει. Συμβαστική G παρακαλώ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, τελική ψηφοφορία τώρα για το σχέδιο γνωμοδότησης. Θα γίνει καταμέτρηση. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Nedlagda. Αποχές. 35 υπέρ. Καμία ψήφος κατά. Καμία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Μογά. Okay. Ωραία. Η δική μου έκθεση τώρα. Κατευθυντήριες γραμμές ε, των πολιτικών απασχόλησης των ε, κρατών μελών. Υπάρχουν δύο τμήματα μέσα στο σχέδιο. Πρώτο τμήμα σε σχέση με τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές, αλλά και μια προφορική ερώτηση και μια πρόταση ψηφίσματος. Θα είναι σύντομος. Για τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές ε, πρόκειται περί της εγκρίσεως των εφισταμένων κατευθυντηρίων γραμμών ε, τριετής διαδικασία για την απασχόληση και για την οικονομία, για όλες δηλαδή τις ενοποιημένες κατευθυντήριες γραμμές. Ε, θα χρειαζόταν κατά τη γνώμη μου ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε τις κατευθυντήρες γραμμές εν ώψη της νέας κατάστασης ως προς την οικονομία και ως προς την κατάσταση της απασχόλησης. Αλλά δεν έχει προκύψει νέα πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κανονικά έπρεπε να είχαν υποβάλει μια πρόταση το Δεκέμβριο ήδη ε, για τη νέα κατάσταση ως προς την απασχόληση και ενδεχομένω ε, σχετικά με τις αλλαγές σε αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές απασχόλησης. Αλλά δεν λάβαμε καμία πρόταση ούτε το Δεκέμβριο ούτε τον Ιανουάριο. Το Φεβρουάριο έφτασε η πρόταση. Τώρα πώς θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία για τις ε, αναθεωρημένες κατευθυντήρες γραμμές. Θα κρατήσει μήνες ολόκληρους. Για να το επεξέλθουμε σε αυτή τη δυσκερή κατάσταση πρέπει να αναλυφθούν σοβαρά μέτρα. Στις κατευθυντήρες γραμμές που υπάρχουν υπάρχει όμως ένα περιθώριο ελιγμών περιθώρια λιγμών για ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ως προς την κατάρτιση παραδείγματο χάρη και άλλες προτεραιότητες αλλά στα πλαίσια των εφισταμένων ε, κατευθυντηρίων γραμμών είτε μιλάμε για την οικονομία είτε μιλάμε για την απασχόληση. Λέω εγώ λοιπόν στην πρότασή μου ότι εγκρίνουμε τις κατευθυντήριες γραμμές και ε, όμως ε, για τον επόμενο χρόνο θέλουμε γέρος να λάβουμε τη νέα πρόταση. Για να προλάβουμε κι εμεί να αποφανθούμε. Να μην επαναληφθεί η ίδια κατάσταση δηλαδή με φέτος. Και πρέπει να έχουμε όλη επίγνωση του ότι έχει αλλάξει άρδινη κατάσταση. Πρέπει να το διαπιστώσουμε αυτό και γι' αυτό υποβάλλουμε προφορική ερώτηση και πρόταση ψηφίσματος. Δηλαδή ταυτόχρονα ε, εγκρίνουμε μεν τις κατευθυντήρες γραμμές, αλλά παρόλα αυτά θέλουμε να τονίσουμε ότι υπάρχει και αυτό το στοιχείο ότι άλλαξε η κατάσταση, έχουμε την οικονομική κρίση, συνδυασμό με το σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας και αλλάζει και η κατάσταση ως προς την απασχόληση. Θέλουμε να τα τονίσουμε αυτά τα στοιχεία. Αυτό είναι το υπόβαθρο, αν θέλετε, τη προφορική ερώτησης και του σχεδίου ψηφίσματος για να τονίσουμε πόσο έκτακτες είναι οι περιστάσεις. Μέσα στην πρόταση ψηφίσματος βασίζομαι σε αυτά που σας έλεγα σε προηγούμενες συνεδρία της Επιτροπής τι, τι πρέπει να κάνουμε δεδομένης της κατάστασης για να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης ε, για να μην αυξηθεί ε, υπερβολικά πολύ η ανεργία. Έξυπνες επενδύσεις, ε, φιλικές προς το περιβάλλον, επένδυση στην κατάρτιση. Αυτή είναι η απάντηση. Επανειλημμένα σας έχω πει ότι ε, στο μέλλον πρέπει οπωσδήποτε να επενδύσουμε στην κατάρτιση. Επ' αυτού πρέπει να συναγωνιστούμε για να αυξήσουμε τις δεξιότητες ε, στην Ευρώπη και να μην ε, αυξάνεται ο αριθμός των ανέργων, αλλά ταυτόχρονα να γίνουμε και πιο ανταγωνιστικοί, αυξάνοντας ε, τις ε, δεξιότητες, επενδύοντας τις νέες δεξιότητες στην Ευρώπη. Αυτά μπορώ να σας πω συνοψίζοντας την έκθεσή μου. Έχω υποβάλει και μία τροπολογία. Ο κύριος Μπούλμαν εξαφανίστηκε τώρα. Θα πάντων έχει υποβάλει διάφορες τροπολογίες που νομίζω ότι ενισχύουν το περιεχόμενο της, του σχεδίου η κυρία Λάμπερτ ε, ε, ήθελε να διαγράψουμε την αναφορά στην αυτοκινητοβιομηχανία. Συμφωνώ, κυρία Λάμπερτ. Δεν θα έπρεπε να κατονομάσουμε μία μόνο βιομηχανία, γιατί η αυτοκινητοβιομηχανία σαφώς αντιμετωπίζει τώρα ιδιαίτερα προβλήματα ε, που αγγίζουν πολλούς κλάδους. Ε, καλό θα ήταν να μην κατονομάσουμε ε, να, μία μόνο βιομηχανία και άρα δέχομαι την τροπολογία της κυρίας Λάμπερτ. Ο κύριος Μπούσελ Μάθιος δέχει έχει υποβάλει δύο τροπολογίες. Τη μία δίχως περαιτέρω μπόρεσα να την υποστηρίξω για την ειδική κατάσταση σχετικά με την άτυπη εργασία των γυναικών και πόσο καλύπτεται αυτό το θέμα ε, δεδομένων των πολιτικών απασχόλησης. Τέλο πάντων την υποστήριξα αυτή την τροπολογία. Για την δεύτερη τώρα τροπολογία ε, είχαμε μία ανακοίνωση Ήρθα σε επαφή με τον ε, κύριο Μπούσελ Μάθιους, του έστειλα mail και δεν μπορώ να συμφωνήσω, εμένω στη θέση μου. Αυτό που ζήσαμε μεταξύ άλλων στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά που ισχύει και σε πολλά άλλα κράτη-μέλη. Δηλαδή, δεδομένες της κατάστασης υπάρχει προφανώς ένας κίνδυνος να ε, χειροτερέψουν συνθήκες εργασίας και να επιδεινωθεί μισθολογική πολιτική θα υπάρχει πίεση προς τα κάτω για τους μισθούς και θα επιδεινωθούν ε, ενδεχομένως και οι συνθήκες εργασίας. Αυτό ήθελα να το τονίσω εγώ στο σχέδιό μου. Στην πρώτη τροπολογία του κυρίου Μπούσελ Μάθιους ε, ήταν προφανές ότι εννοεί πως είναι αναπόφευκτο αυτό δεδομένης κατάστασης, μα δεν συμφωνώ, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό ότι είναι αναπόφευκτο θα πρέπει να προστατεύσουμε και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα το ευρωπαϊκό πρότυπο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι, δεν θα ανταγωνιστούμε, ότι θα ανταγωνιστούμε μόνο με κατώτερους μισθούς και χειρότερες συνθήκες εργασίας. Δεν μπορούμε έτσι να αντιμετωπίσουμε την κρίση στην αγορά. Ακόμη και σε περιόδους κρίσης ε, πρέπει να έχουμε αξιοπρεπείς μισθούς ε, και ε, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Έτσι θα πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Υπέβαλε ο κ. Μπούσελ στη συνέχεια συμβαστική τροπολογία που είναι πολύ πιο ισοσκελισμένη το ομόλογο. Αλλά δεν λέω τόσα πολλά. Δεν εννοούσα ακριβώς αυτό. Εγώ νομίζω πρέπει να μείνουμε στη συλλογική... Λέει ο κ. Μπούσελ ότι θα πρέπει να μείνουμε στις συλλογικές συμβάσεις. Μα ναι, συμφωνώ. Μα το λέω και εγώ στη δική μου τροπολογία. Αλλά ξαναλέω, ε, δεν μπορούμε να μείνουμε ανταγωνιστικοί ε, μειώνοντας ε, τους μισθούς. Δεν μπορώ να αντιδεχτώ την τροπολογία σας. Ναι, να μένουμε στις συλλογικέ συμβάσεις, αλλά πάση θυσία θα πρέπει να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση που θα επιδιώξουμε την ανταγωνιστικότητα μειώνοντα του μισθού. Εμένω στη θέση μου. Ε, η μόνη διαφωνία που έχουμε σε αυτό έγκυται. Κατά τα λοιπά, συμφωνούμε για όλα, όλοι. Κύριε Μπούσελ Μάθιος και ο κύριος Μάν στη συνέχεια. Yes, uh, chairman. Thank you for... Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε να ξεκαθαρίσω τι ήθελα να πω στη δεύτερη τροπολογία. Να ξεκαθαρίσω τι εννοώ. Οπωσδήποτε συμφωνώ μαζί σας. Λέμε δεν θέλουμε να δούμε η γενική αυτή κρίση να μειώσει τους μισθούς και να το εκμεταλλεύεται το κόσμος. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι σε κάποιες εταιρείε οπωσδήποτε στο Ηνωμένο Βασίλειο που υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει, τους δίνεται η επιλογή στου εργαζόμενους. Τους λένε το εξή. τα πράγματα είναι δύσκολα. Ή θα απολύσουμε μερικού ή μπορείτε εθελοντικά να δεχτείτε μείωση του μισθού χ της 100. Ή μερικούς μήνες άδεια με 60% του μισθού διαλέγετε. Επ' αυτές τις συνθήκες έχουν επιλέξει σε κάποιες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι να πληρωθούν λιγότερο από την πολύ χειρότερη επιλογή του να υπάρξουν απολύσεις. Οπότε το να λέμε ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και να λέμε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί μας κάνει να φαινόμαστε λίγο απόμακροι στον κόσμο μας, να μην ξέρουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Οπότε η τροπολογία η δική μου η 7 επί της παραγράφου 14 να πούμε σημειώνει με θλίψη πως είναι αναπόφευκτο πως σε καιρούς οικονομικής κρίσης μπορεί να υπάρξουν κάποιες πιέσεις στους μισθούς προς τα κάτω σε κάποιες εταιρείες ως εναλλακτική λύση στις απολύσεις. Και μετά οπωσδήποτε πρέπει να γίνονται σεβαστές όλες οι συνθήκες, δηλαδή, πρέπει να γνωρίσουμε ότι είναι πραγματικότητα. Για να μην φαινόμαστε και απόμακροι και ότι δεν έχουμε επαφή με την πραγματικότητα. Οπότε αυτή η διατύπωση σας ικανοποιεί. Ο Στίβεν Χιούζ όταν ήταν εδώ είπε πως ε, εάν το έλεγα έτσι θα σας άρεσε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω όμως. Ε, θέλω να ακούσω και τον κύριο Τόμας Μάν και θα σας πω μετά. Also vielleicht schaffen wir es ja, <clears throat> Kompromiss mit jemandem. Ε, τώρα κάνουμε συμβασμό με κάποιον που λείπει από την αίθουσα. Ίσως να έχει και αυτός παρομύστες, αλλά ερχόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό τομέα. Δηλαδή, αν η λύση είναι κάνουμε ανταγωνισμό για ακόμη χαμηλότερους μισθούς, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σωστό είναι αυτό το οποίο είπε ο Φίλιπ, να φροντίσουμε οι εταίροι των συλλογικών συμβάσεων να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους Υπάρχουν τομείς στους οποίους εντάξει μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να, προσμη... να προσπαθήσουμε να επιτρέψουμε μειώσει αλλά μόνο βραχυπρόθεσμα και αλλού υπάρχει αυτό το οποίο έχουμε στην ε, Γερμανία. Δηλαδή οι λεγόμενες ζώνες προστασίας που δίνονται από το κράτος με την δυνατότητα να υπάρξει κάποια εγγύηση ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας. Αυτός μπορεί να είναι ένας όρος, αλλά υπάρχει κλάδους ο οποίος λειτουργεί αυτό το σύστημα και αλλού που δεν λειτουργεί. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικά συστήματα, αυτό είναι σημαντικό. Δεύτερο, εάν μπορούμε να επιτύχουμε τα μέτρα του κράτους που είναι πάντα λεφτά των φορολογουμένων δικά μας να συνδεθούν με όρους και αυτό είναι σωστό. Και δεν μπορούμε να λέμε πώς υποβαθμίζουμε τα πάντα. Γιατί θα οδηγούμαστε συνεχώ σε χαμηλότερου μισθού. σω λοιπόν να μπορούμε να οδηγηθούμε σε κάποιο συμβασμό. Επίση ε, σημαντικό αυτό το οποίο είπε ο Τζιμ Λάμπερτ για την τομέα της βιομηχανία. Είναι ένα τομέα ε, κλείδι, εντάξει, ίσω. Ε, εντάξει, όχι τόσο όσο στη δική μου χώρα, αλλά εξαρτούνται πολλά πράγματα από αυτό. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προμηθευτές, οπότε κλείνω προς αυτό το οποίο είπε ο Γιάν να λέμε πώς πρέπει να παραμείνει αυτό στα κράτη-μέλη, να δουν σε ποιους τομείς θα δώσουν βάρος. Δηλαδή και τρίτον, ήδη προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ποιότητα της εκπαίδευσης των εργαζομένων και χρηματοδοτούμε άτομα τα οποία απασχολούνται με μερική απασχόληση έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε αυτούς τους ανθρώπους να εκπαιδευτούν, να καταρτιστούν για να δουν τι θα κάνουν στο μέλλον όταν θα είναι καλύτερη η κατάσταση, αλλά να έχουν και αυτοί περισσότερα προσόντα. Και να μην γκρινιάζουμε συνέχεια αν δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι εργαζόμενοι κτλ. Γι' αυτό αξίζει να δώσουμε λεφτά για να συνεχιστεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση των εργαζομένων. και λέμε εντάξει ε, μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμο κάτι τέτοιο αλλά έχετε τώρα την ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε αυτό το διάστημα, να εκπαιδευτείτε και μετά να είστε σε μια καλύτερη κατάσταση όταν θα τελειώσει αυτή η κρίση. Δεν θέλω δηλαδή να φύγει αυτό από την, ε, την πολιτική μας ε, ατζέντα και συμφωνώ τελικά με αυτά τα οποία είπε ο Γιάννη. Σας ευχαριστούμε κυρία Λάμπερτ. Ήθελα προφανώς να απαντήσω στον Τόμας Μαν. Ε, μπορούμε να συζητάμε για το εάν η βιομηχανία είναι εξίσου σημαντική, αλλά εδώ μιλάμε για ένα ψήφισμα που αφορά τις ε, κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση. Οπότε όταν μιλάμε για κατευθυντήριες γραμμές, δεν κολλάει αυτό εδώ πέρα. Αν θέλετε να μπει κάπου, ας πάει στο σχέδιο οικονομικής ανάκαψης. Εκεί πάει αυτό το ζήτημα, νομίζω, παρά σε ένα ψήφισμα για τις κατευθυντήριες γραμμές της απασχόλησης. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω λοιπόν στα διάφορα σχόλια. Ναι, κυρία Μωρά, σας δίνω το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα την παρατήρηση που κάνατε λέγοντας ότι θα θέλαμε να έχουμε πραγματικά τον χρόνο για να εμβαθύνουμε στις κατευθυντήριες γραμμές της απασχόλησης. Πέρυσι, θυμάμαι με την Αν Λάνκερ, χρειάστηκε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα σε αυτό το θέμα. το οποίο εμείς προσδίδουμε πολύ μεγαλύτερη σημασία από αυτοί που θέλουν να που δώσουμε εμείς αυτό το θέμα, σε αυτό το θέμα. Έχουμε πολλές εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις που τίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Κατευθυντήριες γραμμές, σχέδιο ανάκαμψης, προσωρινή εργασία, εποχιακή εργασία. Όλα αυτά πρέπει να τα συντονίσουμε διότι Πρόκειται για τους ίδιους στόχους που προασπιζόμεθα εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Αύξηση των ανθρώπινων ικανοτήτων μέσα από την κατάρτιση. Γι' αυτό και εγώ, όπως έλεγε και ο Τόμας Μαν προηγουμένως, συμφωνώ στο πώς, ε, στον τρόπο με τον οποίο συντάξατε την έκθεσή σας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ναι, κυρία Τομασεύσκα. E, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην Πολωνία. Σε μια πόλη της Πολωνίας δέχτηκαν οι εργαζομένοι περικοπή μισθών, αλλά απεδείχθη τελικά ότι και με δεν ήταν δυνατή η καταβολή των, ε, ακόμη και των ε, μειωμένων μισθών και έγιναν ε, διαδηλώσεις. Και πριν από λίγα χρόνια ήταν δύσκολη η κατάσταση. Μειώθηκαν έως και 60% οι μισθοί. Ο κύριος Λουκίνη ανέλαβε τη διεύθυνση του συγκεκριμένου εργοστασίου και ε, απεκλείστηκε ενδεχόμενο να ε, επιστρέψουν οι μισθοί στα προηγούμενα επίπεδά τους. Ε, δηλαδή θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η περικοπή θα γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της κρίσης έκτακτο μέτρο και μετά πρέπει να αυξηθούν και οι μισθοί Και θα πρέπει να επιστραφούν και τα χρήματα που έχουν επενδυθεί στην εταιρεία αφού περάσει η κρίση. Γιατί δεν είναι σωστό οι εργοδότες να, να κερδίζουν και να μην σκέφτονται τους εργαζομένους. Έχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πρέπει αυτά να συνδέονται και με την κρίση. Αυτά νομίζω πρέπει να υποθούν και να υποθούν στεναρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σκομπάρ. Eh, Μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό με τους καιρούς που τρέχουν με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες για τους εργαζομένους να στείλουμε ένα συνενετικό μήνυμα σε αυτή την έκθεση με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμφωνία. Εμείς εδώ θέσαμε δύο στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά και στρεβλώνουν την συνένεση αφορά στη σημασία της αυτοκινητοβιομηχανίας. Θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν θα πρέπει να εξέρουμε ιδιαίτερα την κρίση σε έναν οικονομικό τομέα, διότι όλοι οι οικονομικοί τομείς υποφέρουν. Τώρα στο 14 έχουμε ένα πρόβλημα. Είναι φανερό ότι έχουμε σήμερα δυσκολίες ε, που πλήττουν συγκεκριμένου τύπου επιχειρήσεις. Και θα πρέπει να βρούμε εμεί ένα μέσο παγώματος ε, και διατήρησης ε, των μισθών. Σύμφωνοι. Τα γεγονότα όμως δεν χρειάζεται να τα συζητάμε διότι είναι αυτά τα οποία είναι. Εκείνο το οποίο με ενοχλεί είναι αυτή η πίεση προς τα κάτω των μισθών. Θα έπρεπε λοιπόν να βρούμε μία συμφωνία ώστε το μήνυμα να είναι όσο το δυνατόν πιο, πιο δυνατό. Σας ευχαριστώ. Θα σχολιάσω τις παρατηρήσεις των συναδέλφων ε, αυτά τα θέματα που μας απασχολούν στο ψήφισμα. Λοιπόν, για την αυτοκινητοβιομηχανία, αν θα αναφερθούμε σε αυτή ή όχι, εγώ στη χώρα μου Παίζει πολύ μεγάλο σημαντικό ρόλο η αυτοκινητοβιομηχανία γενικότερα για την οικονομία. Αλλά συμφωνώ με την κυρία Λάμπερτ ε, ότι σε ένα τέτοιο ψήφισμα, παρότι έχει μεγάλο ειδικό βάρος η αυτοκινητοβιομηχανία, δεν πρέπει να αναφερθούμε σε αυτή. Γενικά δεν πρέπει να κατονομάσουμε μία βιομηχανία, έναν κλάδο. Συμφωνώ. Καμία βιομηχανία δεν πρέπει να αναφέρουμε. Τώρα για τους μισθούς, το πάγωμα ή την περικοπή των μισθών για να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης, γνωρίζω ότι σε ορισμένες ε, περιοχές, σε ορισμένες περιπτώσεις συμβαίνει αυτό. Δεν είναι μια γενικευμένη τάση. Αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει να ε, τιμωρούμε ε, κάποιους. Θα πρέπει να εμείνουμε στη γραμμή που χαράξαμε που ανέκαθεν ακολουθούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί ε, με χαμηλότερους μισθούς και χειρότερες συνθήκες εργασίας. Ε, ξέρω ότι έχει γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, γνωρίζω την κατάσταση. Και για αυτή την τροπολογία λέει, τονίζει τη σημασία του να μην αφήσουμε την κρίση να ε, πιέσει προς τα κάτω τους μισθούς και να ε, διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί αυτό και θα κρίνουμε ότι είναι σημαντικό κάθε κράτος μέλος ε, ανάλογα με την εθνική του νομοθεσία και τις πρακτικές να εκπονήσει μια πολιτική ούτως ώστε ο ανταγωνισμός να μην βασίζεται σε μισθούς πείνας στην αγορά. Και επίσης οι συλλογικές συμβάσεις έχουν ευρία εφαρμογή και επίσης ε, ε, γίνεται σεβαστή η ιεραρχία των συλλογικών συμβάσεων και η μισθολογική πολιτική ε, θεσπίζεται μέσα στις συλλογικές συμβάσεις. ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη. Εγώ αυτά είπα, δεν είπα τίποτα παραπάνω. Είναι δύσκολο να μην να αποκλίνουμε από αυτή τη θέση μας ε, που αποτελεί πολιτική συμφωνία. Προσπαθεί να βρει συμβαστική λύση ο κύριος Μπούσελ Λοιπόν, εγώ θα μπορούσα να φανταστώ να πούμε ότι μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά δεν μπορεί να γενικευθεί και να αποτελέσει μια ενός είδου κύρωση για τους εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να ανταγωνιζόμαστε με χαμηλότερους ε, μισθούς ε, και χειρότερες συνθήκες εργασίας. Ε, δεν μπορούμε να πούμε, όπως λέει ο κ. Μπούσερ ότι είναι αναπόφευκτο. Δεν μπορεί να είναι αναπόφευκτο. Εξαρτάται από την πολιτική μας. Αλλά άμα καταφέρουμε, βάση περιπτώσει, να βρούμε συμβαστική ε, λύση, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από την πάγια πολιτική μας. Αυτό έλεγα. Λοιπόν, λίγη συζήτηση και αύριο ψηφίζουμε. Κάτι ξέχασα. Ο καθηγητής Κάλλος Μορέιρο Γκονζάλβες και ο Ρικάρντο Κοντροντρίγκες Κοντρέιρας έχουν συντάξει από κοινού μια έκθεση για τη διαδικασία εφαρμογής των ενοποιημένων κατευθυντηρίων γραμμών. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα Είχαμε απευθύνει επικρίσεις σε σχέση με την ε, συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην εκπόνηση αυτών των ενοποιημένων κατευθυντηρίων γραμμών. Ε, είναι μια ευκαιρία για να ε, εκφράσουμε και εμείς την άποψή μας σε σχέση με αυτή τη διαδικασία. Τώρα, όμως, η νέα διαδικασία θα αρχίσει το 2010. Τώρα θα παραμείνουν οι γραμμές. γραμμέ. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρουμε ακριβώ πώ λειτουργεί η διαδικασία εν ώψη του 2010. Έχετε το λόγο, κύριε Γκονζάλε. Συγγνώμη, συγχωρήστε με, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζομαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε το δικαίωμα υποχρεωτικής διαβούλευσης ε, του Κοινοβουλίου με βάση τη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 128 της ε, Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την έγκριση των κατευθυντηρίων γραμμών απασχόλησης όπως επίσης και το δικαίωμα διαβούλευσης στα πλαίσια της εφαρμογής της στρατηγικής της Λισαβόνας και των πραγματικών προσανατολισμών για την οικονομική πολιτική απειλείται πολύ σοβαρά από την αρχή της συμπλήρωσης του, ε, της συνθήκης του Άμστερνταμ. Για να σας εξηγήσω πώς ε, θα μπορούσε να απαντήσει πολιτικά και τεχνικονομικά το Κοινοβούλιο σε αυτή την ιστορία θα σας ε, εξηγήσω σύντομα. Αν εμείς κάνουμε μία αξιολόγηση της συνθήκης του Άμστερνταμ τα τρία χρόνια από το 2000 μέχρι το 2002 ε, τις ε, προθεσμίες που κράτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να γνωμοδοτήσει για τις πολιτικές απασχόλησης. Διαπιστώνουμε ότι σε αυτή την πρώτη περίοδο, 2000-2002, το Κοινοβούλιο είχε μόνο 1,5 μήνα μπροστά του για να συντάξει την έκθεση. Για το, μεταξύ 2003-2005 μόνο Δύο μήνες είχε στη διάθεσή του το κοινοβούλιο για να εκπονεί στην έκθεσή του. Αλλά όμως με δύο επιβαρυντικά στοιχεία που πρέπει να αναφέρουμε εδώ. Το 2003 στην πρόταση της Κομισιόν ενσωματώνεται και η πρόταση για την υποχρεωτική διαβούλευση για τις πολιτικές απασχόλησης όπως και μη, η, η μη υποχρεωτική διαβούλευση για την οικονομική πολιτική. Αυτό απαιτεί λοιπόν συντονισμό των εργασιών του Κοινοβουλίου και μία τεχνικονομική ε, διεργασία ιδιαίτερα πιο πολύπλοκη. Στις τελευταίες εκλογές ε, το Κοινοβούλιο είχε στη διάθεσή του μόνο δύο εβδομάδες για να εκπονήσει την έκθεσή του. Η κατάσταση δε χειροτερεύει ε, μεταξύ 2006 και 2008 όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το όριο των δύο μηνών για την εκπόνηση της έκθεσης. Αυτή είναι η κατάσταση μας και σήμερα δηλαδή. Αλλά θέλω να το τονίσω, ε, από το 2006 και μετά η Κομισιόν αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού Οπότε η πρόταση για την οποία πρέπει να εκφραστεί το Κοινοβούλιο δεν είναι στρίκτου ένσου ε, αυτό που ορίζεται για την ερμηνεία της συνθήκης στο άρθρο 128 αλλά μία κοινή πρόταση που περιλαμβάνει στο ίδιο πακέτο και την αξιολόγηση για την ε, διεύρυνση της ε, στρατηγικής της Λισαβόνας. Τώρα για, την, τα θέματα της δημοκρατικής νομιμότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για να γνωμοδοτήσετε, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τα εξής. Το χρονοδιάγραμμα της Κομισιόν και αυτός ο τρόπος δια... Ε, μεθόδευσης δεν κάνει διάκριση μεταξύ του 2002 που είχαμε μια στρατηγική, η αλλαγή των κατευθυντηρίων γραμμών και των άλλων ετών όπου η κατάσταση είναι αρκετά επαναληπτική. Και ως νομικός θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρή η κατάσταση ότι η Κομισιόν όταν υποβάλλει την πρότασή της θέτει στο ίδιο επίπεδο το δικαίωμα έκφρασης του Κοινοβουλίου να εκφραστεί βάσει του β του άρθρου 128 της συνθήκης και της διαβούλευσης. Λογικά και με ένα κοινοβούλιο που με τη διεύρυνση αύξησε τα μέλη του και επειδή θα αρχίσει να ισχύει και η συνθήκη της Λισαβόνας, αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ χαμηλή απόδοση σε εκθέσεις του Κοινοβουλίου, σε έναν κορεσμό δηλαδή να οδηγήσει ε, για, ε, ως προς ε, τις ε, γνωμοδοτήσεις του Κοινοβουλίου που πρέπει να δίνονται έγκαιρα δηλαδή πριν από τις συνεδριάσεις των, κλαδικών, των τομεακών υπουργών το Ιούνιο. Η πρόταση έχει ως εξής από πολιτικής πλευράς, ε, διαθεσμικές δηλαδή σχέσεις, για να μπορέσουμε να προσφύγουμε και στο δικαστήριο ε, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η περίοδος, η προεκλογική περίοδος από το Μάιο μέχρι τις θέσεις σε ισχύ της Λισαβόνας η μελέτη προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να πετήσει από την Κομισιόν βάσει του άρθρου 128.2 της συνθήκης να έχει μία προθεσμία πεντάμινη τουλάχιστον για να μπορέσει να εκπονήσει την έκθεσή του. Κυρίως όσον αφορά στην αναθεώρηση των πολιτικών απασχόλησης και μία στρατηγική αρχή του κύκλου. Για τα άλλα δύο χρόνια του κύκλου που είναι απλές αναθεωρήσεις, θεωρούμε ότι με μία περίοδο τριών μηνών όπου δεν θα πρέπει να αλλάξουμε ουσιαστικά το περιεχόμενο των προτάσεων της Κομισιόν, το Κοινοβούλιο θα είχε επαρκή χρόνο στη διάθεσή του. Ο λόγος ε, που ζητούμε αυτή την προθεσμία εκτιμά πέρα δηλαδή από τις εργασίες μετάφρασης που είναι υποχρεωμένες να γίνουν για να μπορούν οι βουλευτές να εργάζονται στις επίσημες γλώσσες αν αρχίσει δηλαδή να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας η αρχή της επικουρικότητας θα απαιτήσει τα εθνικά κοινοβούλια να εκφραστούν κυρίως για τις στρατηγικές αναθεωρήσεις επί του περιεχομένου της Κομισιόν. Υποχρεωτικά λοιπόν απαιτείται να έχουμε μεγαλύτερες προθεσμίες. Τώρα για αυτό το οποίο δεν είναι υποχρεωτική διαβούλευση, δηλαδή οικονομική πολιτική και αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισαβόνας, για τις αρχές ε, του κύκλου ως στρατηγικές, για τις στρατηγικές αναθεωρήσεις θεωρούμε ότι η Κομισιόν πρέπει να παρουσιάζει τις προτάσεις της το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου. Αυτή η στιγμή θα έχει λάβει τους πολιτικούς προσανατολισμούς του Κοινοβουλίου αλλά και για να δώσει χρόνο στο Κοινοβούλιο να παρουσιάσει τη δική του άποψη πριν από το Εαρινό Συμβούλιο. Τώρα, Φόσον αρχίσει να ασχεί η συνθήκη της Λισαβόνας και βάσει του άρθρου 295 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να καλέσει την Κομισιόν και το Συμβούλιο να προχωρήσουν σε μια διαθεσμική συμφωνία για να έχουμε ένα νέο χρονοδιάγραμμα και να ρυθμίσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτό το πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο ένα θέμα περιεχομένου αλλά βάσει αυτού του άρθρου 295 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ένωσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να διεκδικήσει ότι αυτή η διαθεσμική συμφωνία πρέπει να έχει υποχρεωτική, ε, υποχρεωτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση όμως που δεν δεχθεί το Συμβούλιο ή η Κομισιόν είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη λύση, δεν έχουμε άλλη λύση και μιλάμε εδώ για μια περίοδο 2-3 ετών το Ευρωπαϊκό το Κοινοβούλιο να προσφύγει βάσει του άρθρου 232 της ε, συνθήκης της Ευρω... των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να προσφύγει λοιπόν στο δικαστήριο για παράληψη που θα ενίσχυε τη θέση της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. διότι το Κοινοβούλιο μετά από τη συνθήκη του Άμστερνταμ συνεργάζεται με ιδιαίτερη νομιμότητα με το Συμβούλιο και με την Κομισιόν σεβόμενο πάντοτε τις προθεσμίες του. Σε περίπτωση τώρα που το Κοινοβούλιο δεν τύχει τις ίδιες μεταρρύθμισης από το, από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν και άμα λάβουμε υπόψη και την τροποποίηση του 128.2 της συνθήκης, τότε θεωρώ ότι πλήττεται το Κοινοβούλιο και το νόμιμό του δικαίωμα να γνωμοδοτεί. Αυτό λοιπόν θα ενίσχυε την προσφυγή για παράληψη. Επίσης κάτι άλλο το οποίο ορίζεται στη μελέτη είναι τι γίνεται με το 230 άρθρο της συνθήκης δηλαδή προσφυγή προς ακύρωση. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο Υπουργών το Ιούνιο εγκρίνει τις αποφάσεις του, για την απασχόληση χωρίς να έχει αναμείνει στη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου ή εκφραζόμενο ε, σε μία πρόταση της ε, Κομισιόν ε, την οποία θα έπρεπε να είχε εκφράσει το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Γκονζάλες. Δεν είχα διαβάσει εγώ αυτή τη μελέτη, αλλά θα τη διαβάσω. Νομίζω... Αλλά ε, τα έχουμε βιώσει όλοι αυτά, δηλαδή αυτές τις επαφές με το Κοινοβούλιο για τις κατευθυντήριες γραμμές της απασχόλησης. Ε, ε, αποτελούν μια διαδικασία την οποία όμως κανείς δεν έχει πάρει στα σοβαρά από πλευράς Επιτροπής και Συμβουλίου. Έχουμε εργαστεί σκληρά. Συχνά έχουμε πολύ καλές προτάσεις. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Όπως είπε ο κύριος ε, Γκονζάλες, ε, ευγενικά λέμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η θέση μας, αλλά τελικά υπάρχει πρόβλημα γιατί ουδέποτε λήφθη υπόψη η θέση του Κοινοβουλίου. Περιμέναμε τη θέση της Επιτροπής για τις κατευθυντήριες γραμμές. Ε, δεν λάβαμε πρόταση, όπως έλεγα, ούτε το Δεκέμβριο, ούτε τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο μας ήρθε η πρόταση. Επειδή μόνο, μόνο και μόνο επειδή υπάρχει ίσονος κορυφή στο Μάρτιο. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί στα σοβαρά ότι άσκησε επιρροή το Κοινοβούλιο με οποιοδήποτε τρόπο. και αντιδράσαμε με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την πρότασή μου για τις κατευθυντήριες γραμμές. Ε, λέμε ότι θα πρέπει να τις εγκρίνουμε ναι μεν, αλλά να τηρούμε εφ' τις προθεσμίες για τη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο. Πέρα από τα ωραία λόγια, θα πρέπει να είναι και υπόλογη η Επιτροπή, γιατί δεν τη στήρισε τις προθεσμίες. για την επόμενη θητεία, ε, για το επόμενο κοινοβούλιο, ε, είναι σημαντικό να γίνει αξιολόγηση αυτή τη έκθεση, ε, δηλαδή να γίνει αξιολόγηση τη κατάσταση. Ποιε μελέτε θα διεξαχθούν στο ενδιάμεσο διάστημα για τη διαδικασία τη Λισαβόνα και για τι κατευθυντήρε γραμμέ, γιατί θα αντικατασταθούν όλα αυτά από τη νέα διαδικασία θα πρέπει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτή η νέα πολιτική και πρέπει να το διεκδικήσουμε, να διεκδικήσουμε την ουσιαστική συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Να λαμβάνεται υπόψη η άποψη του Κοινοβουλίου και ως προς τη διαδικασία και ως προς τις μακροπρόθεσμες προθεσμίες. Ε, πρέπει να είναι δημοκρατικές οι διαδικασίες εδώ στο Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστούμε πάντως. Ε, στις μελλοντικές του εργασίες ε, το Κοινοβούλιο θα υποφεληθεί από τις εργασίες σας. Και επικυρώνται αυτά που είπα και από την έκθεσή σας, ε, κυρία Φαν Λάνκεν, για κάποιες στρατηγικού χαρακτήρα σκέψεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση για αυτή τη μελέτη. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας πει η μελέτη πού μπορούμε να τη βρούμε γιατί στα πεταχτά την έχω δει και θα ήθελα να διαβάσω με την ησυχία μου. Συμφωνώ πλήρως με την άποψη πως το επόμενο κοινοβούλιο και ελπίζω να συνεχίσουμε και εμείς το κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να, προσπαθ... να συνεχίζει να προσπαθεί να καταλήξει σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο για τα διαδικαστικά γιατί θεωρώ ότι εμείς ως βουλευτές έχουμε μια νομιμότητα όχι μόνο σύμφωνα με το άρθρο 128 της συνθήκης αλλά επειδή είμαστε και αιρετοί από τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματικά πρέπει εμείς να δώσουμε τον ρυθμό και δίνουμε τον σφιγμό του τι γίνεται στις ε, χώρες μας. Οπότε εγώ οπωσδήποτε είμαι υπέρ μιας τέτοιας συμφωνίας. Εγώ δεν θα ήθελα να έχουμε τόσες πολλές ε, δηλώσεις γιατί βλέπω πως οι καθηγητές αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που πηγαίνει πολύ μακρύτερα από τις ε, προθεσμίες εδώ πέρα της Κομισιόν ε, και ένα ζήτημα το οποίο βέβαια τυπικά έπρεπε να το έχουμε συζητήσει πέρσι με τους ε, συναδέλφους και την ε, κυρία Μορέν και κάναμε κάποιες προτάσεις σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Τότε δεν ήταν το πρόβλημα τόσο έντονο ώστε να υπήρχε ανάγκη μια τέτοια έκθεση. Εντάξει, έπρεπε να εργαστούμε γρήγορα, αλλά το πρόβλημα ήταν πως από τυπική σκοπιά το Συμβούλιο κινήθηκε αφού ψήφισε το κοινοβούλιο αλλά δεν αποφάσισε τίποτα βάσει αυτά τα οποία έλεγε το κοινοβούλιο. Αποφάσισε μάλλον πριν ψηφίσει το κοινοβούλιο. Και βεβαίως ε, έπρεπε να βασιστούμε συνθήκη να δούμε ποια είναι τα δικαιώματα του κοινοβουλίου και τελικά αλλά τα τρία θεσμικά όργανα και βεβαίω οι εταίροι του κοινωνικού διαλόγου πρέπει να έχουν την αίσθηση πως όλα τα θεσμικά όργανα είναι σημαντικά για να συνεισφέρουν στη στρατηγική της ε, Λισαβόνας, οπωσδήποτε όσον αφορά αυτές τις ε, κατευθυντήριες γραμμές. Εντάξει, μπορούν να μας βοηθήσουν τα νομικά μέσα και τα δικαιώματα του κοινοβούλιο, αλλά δεν νομίζω τώρα ότι είναι αυτή η σωστή ε, προσέγγιση μας. Δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω. Αν κατάλαβα καλά και ζητώ συγγνώμη γιατί δεν σας είπα, το, το είδα πολύ στα πεταχτά, πως υπάρχει βεβαίως αυτή η υποχρέωση της σύμφωνης γνώμης του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 128 ζητείτε η γνώμη μας αλλά δεν αποτελεί τυπική προϋπόθεση για την τυπική έγκριση αυτού του πράγματος. Αυτό με δυσκολεύει γιατί αυτό το κοινοβούλιο ουσιαστικά καλωσορίζει αυτά τα οποία προέκυψαν από, αυτή την, ε, από αυτές τις τις ολοκληρωμένες ε, κατευθυντήριες γραμμές, γιατί χωρίς μακροοικονομική και μικροοικονομική στρατηγική κτλ. δεν έχουμε δει πολλά πράγματα. Είναι κάτι το οποίο είναι μεμονωμένο και πρέπει να το δούμε σε ένα συνολικότερο πλαίσιο. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να εργαστούμε με δύο προθεσμίες, δηλαδή μία προθεσμία για την υποχρεωτική γνωμοδότηση που μπορεί να είναι πιο μετά και άλλη μία για την διαβούλευση με βάση αυτά τα οποία είχαν προηγηθεί. Τέλος, η τελευταία μου σκέψη προτείνεται πως ε, το Κοινοβούλιο πρέπει να απαιτήσει να έχουμε τουλάχιστον πέντε μήνες για διαβούλευση για τις ε, καθηγητήριες γραμμές. Αυτό όμως σημαίνει τελικά πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταθέσει τις προτάσεις της για τη ολοκληρωμένη αυτή στρατηγική τον Σεπτέμβριο γιατί Υπάρχει ένας μεγάλος νομίζω πολιτικός κανόνας που τον μοιράζομαι και εγώ ότι δεν θα αποφασίσουμε εμείς τον Ιούνιο. Δεν θα αποφασίσει μάλλον το Συμβούλιο τον Ιούνιο γιατί καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να βρει τα εθνικά κοινοβούλια, δεν μπορεί να ψάξει να βρει τους κοινωνικούς εταίρους, να υπάρχει μια συνεισφορά. Πρέπει να γίνει και η μετάφραση και να μεταφερθούν όλα αυτά στα εθνικά σχέδια δράση και είναι και οι διακοπέ, οι καλοκαιρινέ. Οπότε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε το συγκεκριμένο πακέτο αυτό πρέπει να εξηγηθεί και να είναι έτοιμο αρχές της άνοιξης. Ε. Οπότε δεν ξέρω, νομίζω ότι ζητάμε κάπως πολλά πράγματα από την ε, Πρέπει λοιπόν να δούμε, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να γίνουν όλες αυτές οι αξιολογήσεις και να είμαστε έτοιμοι τον Σεπτέμβριο. Εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ για τις ε, προτάσεις σας. Θα είναι οπωσδήποτε πάνω πάνω στα χαρτιά του επομένου Προέδρου. Τη επιτροπή. μα. Ελπίζω να είστε εσεί και να συνεργαστούμε ε, ως Κοινοβούλιο για μια ε, διαθεσμική συμφωνία. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκονσάλε, εφόσον η κυρία Φαν ήθελε να ρωτήσει κάτι για το 2008. Να πω κι εγώ κάτι. Συμφωνώ με την κυρία Φαν ότι αυτό είναι ε, ότι περιπλέκεται ακόμη περισσότερο το θέμα, γιατί τώρα έχουμε εντάξει τις κατευθυντηρίες γραμμές, αλλά στην πράξη ε, θα αποφασιστούν στην Ιαρινή, στο Ιαρινό Συμβούλιο. Δηλαδή, αν και εγκρίνονται τον Ιούνιο, μάλλον επίσημα, οι καθητήριες γραμμές έχουν αποφασιστεί πολύ νωρίτερα. Οπότε ε, έχουμε διάφορες διαδικα... διαφορετικές διαδικασίες ανάλογα αν μιλάμε για τις κατευθυντές γραμμές απασχόληση για την οικονομία και πώς μπορούμε να έχουμε μια ενοποιημένη διαδικασία και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε την επιρροή του Κοινοβουλίου. Πρέπει να αντιληφθούμε δε ότι υπάρχουν και τα εθνικά σχέδια δράσης που πρέπει να αναλυθούν. Να εξεταστούν υπό το φως των προτάσεων. Μόνο μέσα από μια διαθεσμική συμφωνία μπορούμε να διεκπαιρεώσουμε το ζήτημα. Για το 2008 μπορείτε να απαντήσετε κύριε Γκονζάλης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με το κοινό το δίκαιο στο χέρι και υπό τη στενή έννοια του δικαίου μπορεί το κοινοβούλιο να βασιστεί μόνο σε αυτά που λέει η συνθήκη. Διότι εκεί όπου η συνθήκη λέει κάτι δεν είναι το δικαστήριο το οποίο θα αποφανθεί. Και όσες φορές έδωσε δίκιο έδωσε δίκιο στη διεκδίκηση του Κοινοβουλίου για την προσφυγή κατά του δικαιώματος ε, ε; ε επιτρέψτε μου ήταν ιδιαίτερα τσιγκούνικο το, το, δικαστήριο διότι η διαβούλευση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το σχετικό άρθρο και μπορεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Συμβούλιο να αποφασίσει η τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου. Και εδώ είναι τώρα το νομοθετικό πρόβλημα ουσίας. Πώς μπορεί να κερδίσει το Κοινοβούλιο μία νομική μάχη όταν του ζητείτε διαβούλευση γνωμογνώμη για τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Άρα και διαπιστώνουμε και για τη στρατηγική ε, της ε, Λισαβόνας και για τις κατευθυντηρίες γραμμές ε, για την απασχόληση θέλω να καλύψω το κοινοβούλιο. Δεν θέλω να πάει να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το κοινοβούλιο για να χάσει την υπόθεση. Η διαφορά λοιπόν της άποψής μας περιορίζεται εδώ. Σε αυτά τώρα που έκανε η Ευρωβουλευτής έχει απόλυτο δίκιο. Σκοπός είναι να καταλήξουμε σε μια διαθεσμική συμφωνία όπου θα τίθεται επιτάπητο στο πρόβλημα και θα υπάρχει μια πραγματική βούληση των κυβερνήσεων της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου να ξεκινήσουν λογικούς και συμπληρωματικούς κύκλους όπου οι προσανατολισμοί της πολιτικής απασχόλησης θα συμπίπτουν με τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής. Σας ευχαριστούμε. Ναι, το επόμενο κοινοβουλίο θα επιληφθεί του ζητήματος και εγώ συμφωνώ ότι όλα θα ρυθμιστούν στο πλαίσιο μιας διαθεσμικής ε, συμφωνίας. Δεν θα είναι απλό. Είναι απαραίτητο όμως, ε, πρέπει να γίνει από το επόμενο κοινοβούλιο. Για το ερώτημα της κυρίας Φαν για την ερώτηση, υπάρχει σύνοψη της μελέτης που θα σας αποσταλεί αμελητή. Και σε λίγες εβδομάδες ε, θα έχετε ε, την ε, έκθεση. Ολόκληρη την έκθεση. Σας ευχαριστούμε πάντως κύριε Γκονζάλης για τη συνεργασία και για την έκθεση. Λίγη αυτό το θέμα της σημερινής διάταξης και περνάμε στο επόμενο κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων υπεργολαβίας σε αλυσίδες παραγωγής. Ο κύριος Λάσε Λέχτινεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να τονίσω έτσι γρήγορα το υπόβαθρο αυτής της έκθεσης. Συχνά λέγεται εδώ μέσα πως ε, για να λειτουργήσει σωστά η εσωτερική αγορά πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη διασυνοριακή για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το δυναμικό της και βασικά αυτή η έκθεση αυτό ακριβώς αφορά. Με αυτό ακριβώς ασχολείται όπως όλοι ξέρουμε η υπεργολαβία έχει γνωρίσει έκρηξη την τελευταία δεκαετία και αυτό δεν είναι κάτι δυσάρεστο, δημιουργεί οικονομική δραστηριότητα και θέσει εργασία. Χρειαζόμαστε όμως ξεκάθαρους κανόνες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αλλιώ δεν μπορούμε να μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Αγορά Εργασίας που λειτουργεί σωστά. Οι εργαζόμενοι και οι ειλικρινείς εργοδότες ε, ειδικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρώνουν τα σπασμένα της μειονότητας οδήγησαν ακριβώς 8 ε, κράτη-μέλη ήδη να δημιουργήσουν ένα σχέδιο εθνικής αστικής ευθύνης αλλά χρειάζεται μια ευρωπαϊκή λύση για όλη την εσωτερική αγορά εάν είναι πραγματικά να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Συνάδελφοι, ακούσαμε μια εξαιρετική μελέτη από το Ίδρυμα του Δουβλίνου που ασχολούνταν κυρίως με τον τομέα των κατασκευών. Μελέτη η οποία κατέληξε στο ότι οι κανόνες αστικής ευθύνης ε, είναι απαραίτητοι για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους που έχουμε ορίσει. Και μπορώ να πω πως για τη χώρα μου τουλάχιστον πως έχουμε την ίδια εμπειρία κι εμείς η εσωτερική αγορά θα υποφεληθεί από απλούς και ξεκάθαρους κανόνες όχι μόνο για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι αλλά και για να καταπολεμηθεί η μαύρη οικονομία και να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά. Γι' αυτό ελπίζω πως η Επιτροπή μας <coughs> εγκρίνει αυτή την έκθεση στην αυριανή ψηφοφορία. Θα ήθελα εγώ αυτό το θέμα να μην το δούμε ως θέμα αριστεράς δεξιάς στις δύσκολες αυτούς ε, καιρούς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μην έχει τη στήριξη των Ευρωπαίων εργαζομένων και ελπίζω η Κομισιόν να το έχει αυτό κατά νου όταν θα ασχοληθεί ξανά με αυτό το ζήτημα στην επόμενη νομοθετική περίοδο. Χρειαζόμαστε αυτή, αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης γιατί όπως είπα η εμπιστοσύνη προς την Ένωση δεν είναι τόσο μεγάλη μεταξύ των εργαζομένων. Συνάδελφοι, ήθελα να σας ευχαριστήσω και ιδιαίτερα τους κοιόδης σύγητες για τις επικοδομητικές τους τροπολογίες και την καλή συνεργασία. 66 των αριθμών τροπολογίες. Όπως βλέπετε από τον κατάλογο ψηφοφορίας έχουμε μόνο μία ουσιαστική συμβαστική τροπολογία με τους φιλελεύθερους και τους πρασίνους. Δηλαδή η 22 της κυρίας Ρέντερ γίνεται έναν ιωτιμώντας. Ελπίζω λοιπόν να έχω τη στήριξή σας αύριο στην ψηφοφορία για να ωφελήσουμε τους Ευρωπαίους επιχειρηματίες και εργαζόμενους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λετίνεν. Έχουμε τις 66 τροπολογίες και προσπαθήσατε να κάνετε και κάποιες συμβασικές τροπολογίες. Η Γκαμπριέλα Σάνα ζήτησε πρώτο λόγο, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι κύριε Σιγητά. Το φαινόμενο αυτό, το ότι δηλαδή οι εργαζόμενοι δεν τηχάν σωστής μεταχείρισης από τους υπεργολάβους, ε, εργαζόμενοι όπως σας είπα σε υπεργολάβους οπωσδήποτε υφίσταται και πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Κανείς δεν το δέχεται, ούτε και η ομάδα μου. Το θέμα είναι πώς θα το καταπολεμήσουμε. Και εκεί πέρα νομίζω διχάζονται οι απόψεις, εκεί πέρα έχουμε διαφορετικές απόψεις από τον εισηγητή. Και βλέποντας και τις περισσότερες τροπολογίες των σοσιαλιστών και των πρασίνων, ούτε με αυτές νομίζω συμφωνούμε. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποια σημεία για την ε, κοινωνική σφραγίδα που απαιτείται στο σημείο 3. Ωραίο πράγμα. Υπάρχει ήδη στη χώρα μου μια επιχείρηση μπορεί να την κολλήσει αν θέλετε στην πόρτα και να τη σφραγίδα αυτή και να κάνει έτσι, τη διαφήμισή της και πράγματι προσφέρει πολλά πράγματα αλλά κατά την άποψή μου είναι ένα ζήτημα εθνικό και όχι ευρωπαϊκό. Σκεφτείτε μόνο το εξής. Εάν, όπως απαιτείται εδώ πέρα, η κοινωνική αυτή σφραγίδα είναι υπόθεση της Κομισιόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε οπωσδήποτε οι ρήσεις θα θεωρήσουν ότι πάλι έρχονται κανονισμοί από τις Βρυξέλλες και το σημαντικότερο για εμένα προσωπικά, ποιος θα το ελέγξει. Χρειαζόμαστε πάλι τεράστιους μηχανισμούς από την Κομισιόν και τις Βρυξέλλες και στα 27 κράτη-μέλη για το εάν τηρούνται τα κριτήρια ή όχι. Οπότε δεν είναι ζήτημα ε, του ευρωπαϊκού επίπεδου, είναι και του εθνικού. Γι' αυτό είναι για μας αυτό ένα σημείο κλειδί. Δεύτερο, αυτή η αλληλέγγυα ευθύνη που ζητείται σε διάφορα σημεία και θεωρείται εδώ πέρα πανάκια για τις παραβιάσεις αυτές ε, στην αλυσίδα της εργολαβίας και υπεργολαβίας. Η αυτή η κοινή και αλληλέγγυα ευθύνη είναι καλή, αλλά πού είναι η νομική βάση για αυτήν. Ο εισηγητής είπε πως πρέπει να κάνουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωραία αυτά. Αλλά να σας υπενθυμίσω, είμαι και στην Επιτροπή εγώ νομικών υποθέσεων, όπου συζητάμε θέματα και ποινικού και αστικού δικαίου. Ε, μας δεσμεύουν οι συνθήκες. Δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να ζητάμε έτσι, κανονισμούς όσο όμορφοι και αν μας φαίνονται εάν δεν υπάρχει νομική βάση στη συνθήκη. Και αυτό δεν υπάρχει ούτε στις ισχύουσες συνθήκες ούτε συνθήκη της Λισαβόνας δεν υπάρχει τέτοια νομική βάση. Και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι ό,τι θέλουμε να μην το παίρνουμε στα σοβαρά και να απαιτούμε πια πράγματα γιατί μας αρέσουν ή γιατί θα είναι κάτι ευχάριστο να έχουμε έναν ωραίο πανευρωπαϊκό κανονισμό δεν προωθείται έτσι τίποτα και οπωσδήποτε όχι η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν είμαστε τόσο χαλαροί με τη νομική μας βάση δηλαδή αυτή η κοινή και αλληλέγγυα ευθύνη και διορθώστε με αν κάνω λάθος εάν είναι έτσι αν αλλιώς σε άλλες χώρες είναι ζήτημα αστικού δικαίου. Και δεν υπάρχει νομική βάση για κάτι τέτοιο. Έχω σημειώσει κάποια πράγματα για τις τροπολογίες 46 και 51 για το εάν επιτρέπονται. Δεν ξέρω γιατί δεν θα πρέπει να να επιτρέπω, δεν ξέρω προς τι αμφιβολίε. Ίσως ο κύριος Πρόεδρος μπορεί να μας πληροφορήσει τι τρέχει με αυτές τις ε, τροπολογικές ομάδας μας ή μπορεί να το δούμε αύριο. Κάτι ακόμα για την ε, αναφορά που γίνεται στην 38, την τροπολογία, στην πράσινη βίβλο της Κομισιόν για το εργατικό δίκαιο. Μου κάνει εντύπωση πώς ε, αναφέρονται οι σοσιαλιστέ σε αυτή την πράσινη βίβλο. Εγώ ήμουν τυχεροί ως ε, ΕΛΚ ε, να... εγώ θα ήμουν ευτυχής να το παραπέμψετε όλο αυτό το βιβλίο εκεί που ανήκει, δηλαδή στο κάλαθο των αχρήστων. Δεν υπάρχει καμία ασφάλεια εδώ πέρα, είναι το ακριβώς αντίθετο, η ευελιξία με ασφάλεια, αυτό το flexicurity. Δεν είναι αυτό προστασία των εργαζομένων. Ε, προτείνεται επίσης στην 49 την τροπολογία μια μελέτη για ένα νέο κανονισμό για μια ευθύνη η οποία θα προχωρεί παραπάνω στην, στην αλυσίδα. Κοιτάξτε, αν δεν έχουμε νομική βάση δεν χρειάζεται να ζητάμε και μελέτες από την Κομισιόν. Η Κομισιόν έχει τόσες πολλές μελέτες να κάνει, δηλαδή εάν κάνει αυτές ε, τις οποίες ε, νομίμως πρέπει να κάνει και τις κάνει ικανοποιητικά φτάνει, τις περισσεύει δουλειά. Και υπάρχει και μια τροπολογία νομίζω ενό συναδέλφου υπαριθμών 5, ένα εκτιμώντας ε, του κυρίου Κρέμερ που μιλάει για τους μισθούς και τις, όπως ορίζονται και πώς έχει μεταφραστεί εκεί πέρα στα γερμανικά ότι αυτό πρέπει να επαφείται στο πλαίσιο του κάθε κλάδου. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Ώρα μου και στην πλειοψηφία των χωρών αυτό είναι ζήτημα των κοινωνικών εταίρων και των συλλογικών συμβάσεων. Και πολύ καλά ρυθμίζεται εκεί πέρα. Συνοψίζοντα λοιπόν, εμεί ως ομάδα έχουμε σοβαρά προβλήματα με αυτή την έκθεση. Και υπάρχουν κάποια σημεία κλειδιά που ανέφερα που είναι αποφασιστική σημασία για το εάν μπορούμε να υπερψηφίσουμε ή όχι την έκθεση. Δεν πρόκειται, ξαναλέω, για το γεγονός ότι οπωσδήποτε οι καταχρήσεις αυτές ε, όταν έχουμε συμβάσεις εργασίας ε, και υπεργολαβίες πρέπει να καταπολεμούνται. Το ζήτημα είναι μόνο το πώς θα γίνει αυτό και νομίζω εκεί δεν χρειάζεται να πάρουμε ένα πριόνι και να τα κόψουμε όλα στο, στο ίδιο ύψος ή μια μηχανή του γκαζόνου, ό,τι θέλετε. Αλλά παρακαλώ, πρώτα απ' όλα θα αφήσουμε αυτό στους αρμόδιους, στο αρμόδιο επίπεδο, δηλαδή στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Γκαμπριέλα. Μία πληροφορία μπορώ να σας δώσω. Μου λέει η γραμματεία πως κάποιες ε, τροπολογίες δεν επιτρέπονται γιατί συζητούνται στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Ελευθεριών. Κάποια πράγματα τα αντιμετωπίζουν άλλες επιτροπές, οπότε καταθέστε τα εκεί και μπορεί να συζητηθεί εκεί. Μετά έχουμε την Ελίζα Μπέθ Ρέντερ στον κατάλογο των μιλητών. Ναι, ευχαριστώ. Άκουσα αυτά τα οποία είπε η κυρία Στάουνερ με προσοχή. Εν τω μεταξύ βεβαίως το ευρωπαϊκό δίκαιο έχει εξελιχθεί. Μόλις ε, εγκρίναμε την έκθεση Φάβα στην Ολομέλεια όπου το ζήτημα ήταν η συμπεριφορά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Ε, μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου από τον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών. Αν και τελικά η Κομισιόν έκανε μια πρόταση, αρχικά ήταν πρωτοβουλία του Συμβουλίου και εκεί πέρα περιέχεται αυτό το οποίο γράφει ο συνάλφος Λέχτινεν. Αυτό αποφασίστηκε. Οπότε λογική συνέπεια νομίζω είναι να αναφέρεται σε αυτά και να προχωρεί, να εξελίσσει αυτή τη σκέψη και να κάνει προτάσεις. Οπότε θεωρώ αυτά τα οποία... Δεν μπορώ να παρακολουθήσω αυτά τα οποία είπε η κυρία Στάουνερ. Το Συμβούλιο, δηλαδή τα κράτη-μέλη στα οποία αναφέρθηκε η συνάδελφος ε, από κοινού με την Κομισιόν ε, θεωρούν πως πρέπει να υπάρξει εδώ πέρα μια περαιτέρω εξέλιξη και δημιούργησαν με αυτόν τον τρόπο μια βάση πάνω στην οποία πατάει η έκθεση Λέχτινεν. Οπότε αυτό το οποίο λέει η κυρία Στάουνερ δεν ισχύει. Έχουν αλλάξει γραμμή οι πλεύσεις στα κράτη-μέλη. Οπότε εμείς υποστηρίζουμε και την έκθεση. Ευχαριστούμε κυρία Σρέντα. Ο Γιάν Κρέμερ, ο οποίος προφανώς ε, μας παρακολουθεί με αγωνία. Ευχαριστώ, Τόμας. Θα μιλήσω λίγο στα γερμανικά γιατί υπάρχει ένα μεταφραστικό λάθος ε, στην ε, τροπολογία 5. Η πρότασή μου εκεί ε, αναφέρεται λέει ότι ακολούθως άρα και τα λοιπά, αλλά δεν, είναι, δεν συμφωνεί με το αγγλικό κείμενο. Θα προσπαθήσω να το δω με τη γραμματεία, γιατί ε, εκεί πέρα γράφει κάτι άλλο από αυτό το οποίο εγώ εννοούσα, περιπτώσει. Αυτό το συνεπώς δηλαδή. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω επειδή έχω ψάξει τα τελευταία χρόνια αυτό το τομέα ακριβώς τα κατώτερα στρώματα αυτής της ε, αλυσίδας αν θέλετε δεν τηρούνται οι συνθήκες εργασίας οι προβλεπόμενες γιατί ακριβώς μιλάμε για μαύρη εργασία για το χύψη πράγμα και είναι συνήθις πρακτική και υπάρχει, ξέρετε και στη Γερμανία, η αποφυγή των συλλογικών συμβάσεων εργασία. Γι' αυτό ακριβώς έχω κάνει και αυτή την ε, τροπολογία. Ευχαριστώ Γιάν. Ε, πράγματι είναι μεγάλο πλεονέκτημα η πολυγλωσία και σε συγχαίρω. Ο Λουίτζι κατόπιν έχει το λόγο. No, σε μένα αναφερόταν αλήθεια. Λοιπόν, εγώ ήθελα να υπογραμμίσω από τη συζήτηση που ακούσαμε να περιφρουρήσουμε το θέμα της υπερβολαβίας ούτως ώστε να αποφύγουμε τις καταχρήσεις. Η υπεργολαβία έχει μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή οι επιχειρήσεις με τομεακές εργασίες εχμής να παρεμβαίνουν στην υπεργολαβία της ε, ε, βασικής επιχείρησης και βελτιώνουμε έτσι την ε, παραγωγική αλυσίδα. Και δεν θέλουμε οι υπεργολαβία να χρησιμοποιείται με τρόπο κατάλληλο παραβιάζοντας κανόνες όχι μόνο μισθοδοτικούς αλλά να αποφύγουμε ένα μισθολογικό ντάμπινγκ αλλά και ντάμπινγκ άλλων κανόνων όπως είναι υγεία, ασφάλεια στο χώρο της εργασίας δηλαδή η βασική επιχείρηση που κέρδισε τη δημοπρασία έχει δεσμευτεί για ορισμένες ε, συνθήκες δίνοντας όμως την υπεργολαβία και μόνο με την ευθύνη του υπεργολάβου μπορεί να οδηγήσει στην παραβίωση αυτών των κανόνων. Δεν είναι το στόχος που μας διασπά εδώ, είναι το θέμα των αρμοδιοτήτων. Εγώ θυμίζω ότι η κοινοτική διάσταση ήδη έχει παρέμβει με διάφορες ε, οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της υπεργολαβίας. Αλλά γιατί αυτό. Υπάρχουν κανόνες που αφορούν στη λειτουργία της κοινή αγοράς, της ενιαίας αγοράς και η ευρωπαϊκή διάσταση θέλησε να μην μπορέσουμε να παραβιάζουμε, να στρεβλώνουμε αυτούς ε, τους στόχους ε, κατά την υπεργολαβία. Δεν μπορούμε εμείς σε μία ε, δημοπρασία να χρησιμοποιούμε όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διότι θα ήταν παράνομο όταν θέλουμε εμείς να προωθήσουμε την ενιαία αγορά να έχουμε τέτοιου είδους πολιτικές. Είναι δυνατόν εμείς χρησιμοποιώντας αυτή την ίδια πολιτική βάση στην κοινοτική τους διάσταση να αγνοούμε ορισμένους κανόνες που σημαίνουν ε, βασική ευθύνη διότι όταν εγώ ως βασική κύριε εταιρεία δίνω την εφαρμογή στον ε, μεταπράτη τότε θα σεβαστώ, θα πρέπει και εγώ να δεχθώ τους κανόνες σεβασμού των εθνικών πρακτικών. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η νομική βάση υπάρχει, διότι δεν είναι δυνατόν να φανταστούμε ότι υπάρχει για την υπεράσπιση της ενιαίας αγοράς και να μην υπάρχει στην προκειμένη περίπτωση. Διότι αυτό το οποίο θέλουμε είναι να χρησιμοποιούμε την υπεργολαβία, γιατί μπαίνει στην παραγωγική διαδικασία και αλλά να μην το χρησιμοποιούμε ως ε, άμεση ε, απειλή και ο συμβιβασμός όπου έχουμε σχετικά από μία συνάδελφο είναι πολύ καλός και φυσικά θα περάσω από το σπίτι αλλά σας ε, δίνω το πλαίσιο της αρμοδιότητας των κρατών μελών που δεν παραβιάζει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Εγώ ελπίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν συμβιβασμό και η πράσινη βίβλος που ασχολιόταν με την Flexi ε, ε, Security ε, αντιμετώπιζε και το θέμα της υπεργολαβίας. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ πιο σημαντική παρατήρηση στο προηγούμενο σημείο. Ευχαριστώ Λουίτζι. Και η Άννα Φαλανκέρη, η οποία υποσχέθηκε ότι θα μιλήσει πολύ λίγο. Ευχαριστώ. Δεν θα βγάλω εγώ τώρα λόγο για την σημασία της πολιτικής μας για την ευθύνη σε ολόκληρη την αλυσίδα απλά για τα επιχειρήματα που ακούστηκαν περί της νομικής βάσης να υπενθυμίσω στην κυρία Στάουνερ πως υπάρχει νομική βάση και μάλιστα ενέκρινε την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια οδηγία για τις κυρώσεις στους εργοδότες οι οποίοι απασχολούν ε, ανθρώπους ε, χωρίς χαρτιά, εν πάση παρανόμους. Οπότε είναι λίγο κοινικό να λέμε πως ε, δεν ισχύουν οι κανόνες ε, τους οποίους εγκρίναμε γιατί αφορά μόνο την ε, πρώτη, το πρώτο επίπεδο αν θέλετε και δεν κοιτάμε παρακάτω στην αλυσίδα. Ήδη η Κομισιόν ήρθε με μια πρόταση για μια ευθύνη σε ολόκληρο το μήκος της αλυσίδας. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να λέμε πως δεν υπάρχει νομική βάση για μια τέτοια κοινωτική πρωτοβουλία. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Λάσε, έχεις το λόγο. Δεν υπάρχει κανένα από την Επιτροπή, από ό,τι μου είπαν. Δεν χρειάζεται για τους τροπολογίες, έτσι δεν είναι. Την περασμένη φορά ακούσαμε κάποιον από την Επιτροπή. Λάσε. Πρόεδρε, σύντομα θα πω επί της αρχής, αν έχουμε διασυνοριακά προβλήματα, οφείλουμε να έχουμε και διασυνοριακές λύσεις. Οπότε, σας παραπέμπω τροπολογία 49, με λίγη καλή θέληση, δεν μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι αντιβαίνει στις επιθυμίες ε, της κυρίας Τάουνερ, του κυρίου Κωσιλόβου, γιατί ζητάμε απλά από την Επιτροπή να δράσει, να αρχίσει να κάνει κάτι ε, για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστούμε. Αύριο θα ψηφίσουμε στις 9. Μην ξεχάσετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες. θα είναι, γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έχουμε και αρκετές εκθέσεις. Επόμενο σημείο 7. Σάμπα Σόγκορ. Πολυγλωσία. Πλεονέκτημα για την Ευρώπη. Έχετε το λόγο. Uh, ναι, θα μιλήσω αγγλικά. Η πολυγλωσία δεν είναι μόνο μια δυνατότητα για την εκμάθηση γλωσσών, αλλά όπως λέει και ο νέος τίτλος, είναι πλεονέκτημα στο σχέδιο γνωμοδότησης. Αυτό, αυτή τη γραμμή ακολουθώ. Ένα κεφάλαιο αποτελεί η πολυγλωσία για όσους θέλουν να εργαστούν και ως ε, μέλος της Επιτροπής Απασχόλης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλες τις τροπολογίες σας. Βέβαια κάποιες ήταν εκπρόθεσμες, κάποιες έπρεπε κανονικά να υποβληθούν στην Επιτροπή Πολιτισμού. Στις περισσότερες περιπτώσεις θα τα καταφέρουμε να βρούμε συμβαστική λύση. Περιμένω τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε Κούστα, ε, ο πρώτος στον κατάλογο μιλητών. Ε, εντάξει, θα βιαστεί λίγο ο εισηγητή. Θα περιοριστώ σε δύο ζητήματα. Με ικανοποιεί η πρόταση της Ρίας Ιουμεν Ρόιτεν και της Καβριέλας πως πρέπει να μαθαίνουμε όχι μόνο αγγλικά αλλά και τις γλώσσες των γειτόνων μας και αν μάθουμε πολύ γρήγορα τα αγγλικά υπάρχει ο κίνδυνος οι γείτονες να επικοινωνούν μόνο στα αγγλικά και να μην γνωρίζουν τις ε, γλώσσες των γειτόνων τους και με ευχαριστεί το ότι είναι αυτό εδώ μας και μετά για την δική μου τροπολογία που έχει τον αριθμό 14 κυρίως γιατί άκουσα πως ε, συγητής, ο κύριος Σόγκορ έχει κάποιες αμφιβολίες θα ήθελα να την αιτιολογήσω λίγο Οι ερευνητές μας λένε ξεκάθαρα πως ε, η μητρική γλώσσα είναι σημαντική για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών και για τους μετανάστες είναι σημαντικό να την μάθουν εκεί που έχουν τις βαθικές τους ικανότητες. Για οπότε εγώ δεν λέω με τροπολογία αυτή να λέω να πω πως ε, καλύτερα οι μετανάστες να μάθουν τη δική τους γλώσσα και να περιφερειοποιηθούν και να μην ενσωματωθούν αντίθετα. Για να μάθουν καλύτερα τη γλώσσα της χώρας στην οποία βρίσκονται πρέπει να ξέρουν και την δική τους, τη μητρική τους καλά. Ε, το αναφέρω γιατί εδώ πέρα οι συντονιστές ε, γνωρίζουν πως εργάζομαι χρόνια εδώ πέρα και δίνω βάρος ε, στον τομέα αυτών της ενσωμάτωσης, απλά πρόκειται για ένα επιστημονικό δεδομένο. Και αν το αγνοούμε αυτό, δυσκολεύουμε την πρόσβαση των ανθρώπων αυτών στις δικές μας ε, γλώσσες. Γι' αυτό, κύριε Σόγκορ, θα ήθελα να ξαναδείτε την ε, τροπολογία 14 και ίσως να την υποστηρίξετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πράγματι υπενθύμηση και στους Άγγλους αυτό ε, να κάνουν μια προσπάθεια για καμία άλλη γλώσσα πριν των Αγγλικών. Κυρία Κωτή έχει τον λόγο. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω την επιχειρηματολογία που ανέπτυξα την περασμένη φορά. Θέλω να ευχαριστήσω ενθέρμως τον εισηγητή και τους συνεργάτες του. Έχουμε βρει πολύ καλές συμβαστικές λύσεις ε, και νομίζω ότι διασαφηνίζουμε έτσι και την έκθεση, ε, την γνωμοδότηση μάλλον και την καθιστούμε πιο συγκεκριμένη. Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο, τον κύριο Γκούστας, ε, η μητρική μας γλώσσα είναι που μας παρέχει τις βασικές γραμματικές δομές που μας επιτρέπουν να μάθουμε ξένες γλώσσες. Αυτό έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Δεν γίνεται αν δεν κατέχει κάποιο τη μητρική του να μάθει ε, ξένες γλώσσες. Πρέπει πρώτα να κατέχει κάποιος πλήρως την μητρική του γλώσσα. Εμείς θα θέλαμε να υποστηρίξουμε την τροπολογία 14. Αν ε, δεχτεί ο εισηγητή να το σκεφτεί περαιτέρω, πολύ θα μας ικανοποιούσε. Δεν νομίζω ότι δημιουργεί τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτή η τροπολογία. Ε, ναι, ευχαριστώ. Κοιτάξτε για αυτό το οποίο είπατε για την τροπολογία 14. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά το σκέφτηκα και με άλλες τροπολογίες πως ε, δεν είναι θέμα της δικής μας Επιτροπής αλλά της Επιτροπής Πολιτισμού να δεχτεί αυτή την τροπολογία. Εγώ δεν έχω αντίρρηση πάντως. Είναι σαφές. ως μέλος μιας μεγάλης ε, μειοψηφίας προσπαθώ να περιοριστώ στις τροπολογίες της δικές μας ε, υποτροπής. Κανείς δεν μπορεί να πει πως, ε, πως δεν είμαι αμερόληπτος. Απλά νομίζω πως αυτό πράγματι πάει στην Επιτροπή Πολιτισμού. Σας ευχαριστώ. Άλλος ομιλητής δεν υπάρχει για αυτό το σημείο. Λίγη συζήτηση και αυτή την γνωμοδότηση θα την ψηφίσουμε αύριο. Πάμε τώρα στα δικαιώματα των ασθενών στην διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Ο κύριος Μπραγκέτο. io ho già fatto conoscere ovviamente le proposte di... Γνωρίζετε ήδη τις συμβαστικές προτάσεις. 8-9 το αριθμό. Όσο και το πλήστον, ο στόχος αυτών των συμβαστικών τροπολογιών είναι να εμπλουτίσουν την έκθεση και συμπεριλαμβάνει τι προτάσει των συναδέλφων. Υπάρχουν δύο συμβαστικέ τροπολογίε που λίγο μα δυσκολεύουν. Οι συμβαστικέ ε και F. Για το άρθρο 8 και οι δύο. για την νοσοκομιακή περίθαλψη και τις ειδικές ε, νοσηλευτικές υπηρεσίες καθώς και ε, τον κατάλογο το, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, δηλαδή οι αρμοδιότητες που αναφέρονται εκεί αποδίδονται στα κράτη-μέλη και η ε, παράγραφος 3 φέρει επί της ε, πρώτερης έγκρισης που χρειάζεται, χρησιμοποιείται ένα μόνο κριτήριο, το κράτος μέλος προορισμού πρέπει να προβλέψει ένα σύστημα πρώτερης έγκρισης ε, σε περιπτώσεις όπου ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα η κινητικότητα των ασθενών για την παροχή των ε, υγειονομικών υπηρεσιών ή για την ε, χρηματοοικονομική ισορροπία του κράτους. Αυτές είναι οι πιο δύσκολες συμβαστικές τροπολογίες, αν θέλετε που τροποποιούν την ε, πρόταση της ε, Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι υπόλοιπε απλώς εμπλουτίζουν την έκθεση γιατί και λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λίν και η κυρία, ε, συγγνώμη, η κυρία Λίν και η κυρία Φανλάγκεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την συνεργασία του. Ξέρω ότι δεν θα υποστηρίξετε την 154 τροπολογία μου γιατί καλύπτεται βέβαια από τη συμβαστική τροπολογία. Χαίρομαι που ως επιτοπλίστων καλύψατε τα στοιχεία της τροπολογίας 154 αλλά έχω ακόμη έναν ανησυχία για τα 191. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν ενεργητικά τα ΜΕΤΑΔΗ σχετικά με τη, ε, τους επαγγελματίες, ε, σχετικά με επιθαρχικά μέτρα κατά της δυνατότητάς τους για εγγραφή ε, στο ιατρικό σώμα ή στη, για την παροχή υπηρεσιών. για ένα κράτος μέλος είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας ασθενής να ξέρει ότι θα ε, ακολουθεί στην αγωγή με έναν ε, γιατρό που έχει έρθει από ένα άλλο κράτος μέσα, αλλά πρέπει να ξέρει αν έχει διαγραφεί από τον Ιατρικό Σύλλογο. Ε, και έχουμε και την, το ψήφισμα από 15 Μαρτίου 2007 για την κοινοτική δράση σχετικά με την παροχή, διασυνοριακή παροχή και νομικής περίθαλψης. Γιατί λοιπόν είστε κατά τις 191 εφόσον προστατεύουμε τους ασθενείς ε, για να ε, εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ε, θεραπεύονται από έναν επαγγελματία ενώ δεν θα έπρεπε γιατί έχουν διαγραφεί από τον ιατρικό σύλλογο ενός άλλου κράτους μέλους. Τέλος πάντων ευχαριστούμε για τη συνεργασία και ευχαριστώ που εγκρίνατε τόσες πολλές από τις τροπολογίες μου και που συνεργαστήκατε μαζί μου για τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Φανλάνκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε που μιλάω αγγλικά μετά την έκθεση για την πολυγλωσία, αλλά όπως ξέρετε είχαμε συνεδρίαση της ομάδας και επειδή οι συνάδελφοι δεν ε, καταλαβαίνουν αγγλικά, έχω τις σημειώσεις μου, δεν καταλαβαίνω ολλανδικά, έχω τις σημειώσεις μου στα αγγλικά και ζητώ συγγνώμη και του διερμηνείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τους καλούς συμβάσμους. Νομίζω ότι ξεκαθαρίσαμε αρκετά πράγματα, αλλά υπάρχουν ακόμα κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Πρώτα απ' όλα, να επισημάνω συναδέλφους πως καταφέραμε να ορίσουμε το πεδίο εφαρμογής αυτό, αυτής της οδηγίας. Μιλάμε για κινητικότητα μόνο ασθενών και όχι επαγγελματιών της υγείας. Κανείς δεν μας λέει πως είναι δηλαδή Μπολκενστάιν Β. Είναι μόνο για την κινητικότητα των ασθενών. Το άλλο πρόβλημα. Όταν περνάμε αυτή τη γραμμή πρέπει να υπερψηφίσουμε και την τροπολογία 37 των πρασίνων και την 48 των πρασίνων που περιορίζουν την έννοια της διασυνοριακής υγειονομικής περιθέλψης μόνο στους ασθενείς και όχι στους επαγγελματίες της υγείας. Μπορείτε να πείτε πως είναι μόνο τα εκτιμώντας, αλλά τα εκτιμώντας πρέπει να συνάδουν και να συμφωνούν με τα άρθρα. Δεύτερον, συμφωνούμε όλοι νομίζω πως πρέπει να εισαχθεί εδώ πέρα μια σαφής ρήτρα που θα δίνει προτεραιότητα στον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και να διαγράψουμε τα υπόλοιπα γιατί είναι πολύ ε, περίεργα. Αυτό γίνεται πολύ σωστά στην τροπολογία 73 των πρασίνων. Ακόμη καλύτερα και από τη δική μου την 71. Γιατί οι πράσινοι λένε ξεκάθαρα πως εάν υπάρχει κάποια σύγκρουση ο κανονισμός προηγείται κατησχεί. Ξέρω πως θέλει ο εισηγητής να υποστηρίξει τη δική μου την 72 τροπολογία της ε, Ομεν αλλά θέλω να σκεφτεί ο εισηγητής μήπως ε, αυτό η παραπομπή δηλαδή που κάνει η Ρία στον κανονισμό 883 τον καινούριο δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς στον 74 ε, οπότε μπορεί να υποστηρίξει είτε τη δική μου την 71 είτε την 73 των Πρασίνων. Εγώ προτιμώ την 73 εν πάση Τρίτον, νομίζω πως ε, προσπαθήσαμε και καταφέραμε να περιορίσουμε τον ορισμό της υγειονομικής περίθαλψης σε αυτά τα οποία καλύπτονται από τα κράτη-μέλη. Και ευχαριστώ τον συγγητή που υποστηρίζει την 76 των Πρασίνων που είναι καλύτερη από τη δική μου. Γιατί εγώ στη δική μου εξακολουθώ να αναφέρομαι στους επαγγελματίες υγεία και ξέρετε τι συζήτηση είχε προκαλέσει αυτό. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την υποστήριξη των τέταρτων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αναγνωρίζουμε πως η πρώτερη έγκριση είναι ο γενικός κανόνας και όχι η εξαίρεση. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ορίσουν τι είναι νοσοκομιακή και ειδικευμένη περίθαλψη και ευχαριστώ τον εισηγητή. Η πρώτερη περίθαλψη το σύστημα αυτό είναι σημαντικό μέσο για να μην γίνει κινητικότητα των ασθενών ε, κάτι το οποίο θα επηρεάσει πάρα πολύ τα εθνικά τη μελη ε, Επίσης έχει προσθεθεί μια τελευταία πρόταση και κάποιοι τρόμαξαν. Αλλά η τελευταία αυτή πρόταση ε, δεν είναι παρά σύνθεση των όρων του άρθρου 3 της παραγράφου 8 α και β, 1 και 2 και ποιοι είναι μάλιστα ευρύτερα διατυπωμένοι, οπότε διευρύνει τις περιπτώσεις στι οποίε μπορούν τα κράτη-μέλη να βασιστούν στην πρώτη εξοδότηση. Όπως σας είπα γίνεται ο κανόνας και όπως είπε και ο εισηγητή, πρόκειται για τη συμβιβαστική τροπολογία κλειδί όπου α και F, όπου περιορίζουμε σαφώς το πεδίο εφαρμογής οδηγίας. Σημαντικό επίσης είναι ότι ο εισηγητής μας αποδέχτηκε τις προτάσεις μας όχι μόνο να δούμε τις εκροές ασθενών αλλά και τις εισρωές. Οπότε σας ευχαριστώ και για τον συμβασμό επαριθμών G. Το μόνο το οποίο δεν είναι συνεπές με τα υπόλοιπα και είναι σημαντικό για την ομάδα μου είναι η προτινόμενη νομική βάση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι το άρθρο 95 περί ολοκλήρωσης εσωτερικής αγοράς. Είναι η μόνη υπαρκτή νομική βάση για να πατήσουμε. Αλλά εδώ πέρα μας δίνεται η ψευδέστηση πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη διασυνοριακή υγειονομική περιθλίψη μόνο με μέσα εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε, η ομάδα μου επιμένει, να έχουμε βεβαίως το άρθρο 95 που το χρειαζόμαστε αλλά να αναφερθούμε και στο άρθρο 152 περί δημόσιας υγείας και το 106 περί συμφωνίας ε, περί υπηρεσιών με συγχωρείτε, γενικού δημοσίου συμφέροντος ε, κοινή οφειλίας για να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για τη δημόσια υγεία και την κοινωνία κτλ. Αυτά ήταν τα σχόλιά μου κύριε Πρόεδρε. Αυτά άμα ξεκαθαρίσουμε και τα κάνουμε σωστά, ως Επιτροπή Απασχόλησης θα έχουμε δώσει ένα σαφές μήνυμα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, αλλά και πάλι θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα που κάνω συνέχεια. Είναι σαφής οι αρμοδιότητες της Επιτροπής μας, γιατί κύριε Πρόεδρε και κύριε Σιγητά, μπορεί να είναι ξεκάθαρο πως σε αυτή την Επιτροπή είμαστε ικανοί να καταλήξουμε σε καλό αποτέλεσμα, αλλά εάν αυτό το αποτέλεσμα μετά δεν υιοθετείται, ε, λόγω αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή Περιβάλλοντος δεν έχουμε καμία διαβεβαίωση. Ε, το ξαναλέω και το ξαναλέω αυτό το ζήτημα γιατί για την ομάδα μου είναι θέμα κλειδί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα το σχολιάσω αργότερα. Η κυρία Ούμεν Ρόιτεν και η κυρία Λάμπερτ ακολουθούν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εχθές ε, είχα την ευκαιρία να συζητήσω επί μακρόν με τον συνάδελφο Μπραγκέτο για αυτό το θέμα και ήθελα να συζητήσω και με την Άννα Φανλάκεν, αλλά εντάξει έχουμε χρόνο ακόμη να το συζητήσουμε. Να σας πω τι έγινε με τις 72 και 74. Ε, η μία έχει σχέση με την περίοδο πριν από τη θέση εφαρμογή και η 74 για με την περίοδο μετά τη θέση εφαρμογή. Θα σας το εξηγήσω και καλύτερα. Έχουμε πάντως πολλούς ενδιασμούς για την ελεύθερη κυκλοφορία των καταναλωτών στον τομέα της υγείας πολύ περισσότερους συνδυασμούς ε, από ότι το ΔΕΚ παραδείγματος χάρη και θεωρώ ότι ε, θα μπορέσω να συμπαραταχθώ με την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλλον παρά με διάφορες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Εγώ θέλω να είμαι ρεαλίστρια, Πρόεδρε. Ε, θέλω να ε, επιδιώκουμε κάτι που μπορούμε να επιτύχουμε όταν υποβάλλουμε συμβαστικές τροπολογίες. Στο άρθρο 8 λοιπόν... Ε, έχουμε μια σειρά από διατάξεις που αποπειράθηκαν να τροποποιήσουν οι συνάδελφοί μου και βλέπω ότι προσπαθούμε να αφαιρέσουμε αρμοδιότητες από την Επιτροπή. Διότι η Κομισιόν δεν είναι σε θέση να ορίζει πότε ένας ασθενής μπορεί να περνάει τα σύνορα και πώς ορίζεται η θεραπεία και πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε όλα αυτά και τα κέντρα αριστείας Διότι αν δεν γίνει αυτή η συμπερίληψη δεν θα έχουμε ποτέ μα ποτέ ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών. Και στην επόμενη εκλογική, ε, προεκλογική εκστρατεία εγώ θα θέσω ως πρώτο μου στόχο την κινητικότητα των ασθενών. Και πιστεύω ότι όλα εδώ όσα υποβάλλονται ως προτάσεις είναι πάρα πολύ συγκρατημένα. Εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον των κρατών μελών που θέλουν να επηρεάσουν τους ασθενείς κατά την είσοδο στη χώρα. Δεν έχω τίποτα εναντίον. Αλλά άμα όλα αυτά γίνονται με 27 διαφορετικούς τρόπους, τότε από την οδηγία δεν υπάρχει πλέον τίποτα. Θα πρέπει λοιπόν οι συνάδελφοι να βρεθούν γύρω από ένα τραπέζι και να κοιτάξουμε να βρούμε έναν κοινό παρανομαστή διότι έχουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρόκειται εδώ για κωδικοποίηση μίας απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εδώ πρόκειται για κάτι το οποίο πέτυχαν μερικοί πολύ γενναίοι πολίτες και το κατέκτησαν μέσα από το δικαστήριο. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε πολύ συγκρατημένοι ως προς το μέτρο αυτό. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συγγετή και εγώ με τη σειρά μου για τη δουλειά που έκανε Συμφωνώ απολύτω με την Αν Φαν που απευθύνει έκκληση προ του συναδέλφου να υπερψηφίσουν τι τροπολογίε των ε, πρασίνων. Ε, αλλά αυτό δεν σα ξαφνιάζει. Συνήθω ε, συμφωνούμε από αυτό. Επίση, για μία από τις τροπολογίες με καθησύχασε γιατί είχα κάποιες απορίες. Σε σχέση με αυτά που είπε η Ρία και άλλοι, σε αυτή τη συζήτηση. Θα ήθελα να πω το εξή. Ε, επειδή έχουμε εδώ μια ισορροπία, δηλαδή θέλουμε συνθήκε αγορά, θέλουμε οι ασθενεί να επιλέγουν πού θα πάνε για την περίθαλψή του ε, και άρα φυσικά είναι ξεκάθαρα ευθύνη των κρατών μελών η παροχή των ε, υγειονομικών υπηρεσιών, γενικότερα υπηρεσιών κοινή ωφέλεια. Θα Ήθελα ξεκάθαρα μέσα στο διατακτικό και όχι μόνο στα εκτιμώντα, όχι μόνο στην αιτιολογική έκθεση, στο διατακτικό νομικό πώ να συνδέονται αυτά με τα άρθρα 152 και 16 να υπάρχει μια ισορροπία και ξαναλέω μέσα στο διατακτικό όχι μόνο στα εκτιμώντας γιατί ξέρετε ότι δεν έχουν βάρος τα εκτιμώντα ε, μιας οδηγίας ε, ενώπιον του ΔΕΚ για την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής ε, από, από πλευρά των ασθενών ε, να διατρέξουν του κινδύνους που θέλουν και να δώσουν τα λεφτά τους εκεί που θέλουν εντάξει αλλά τώρα η αποζημίωση βάσει του εθνικού συστήματος ε, είναι ένα άλλο θέμα δηλαδή πρέπει να υπάρχει ασφάλεια σχετικά με το αν θα υπάρξει αποζημίωση των εξόδων ναι ή όχι αν θέλουμε πλήρη ασφάλεια τότε η πρώτερη έγκριση ε, έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί αν δεν έχετε ένα τέτοιο σύστημα πρώτερη έγκριση, ελοχεύει ο κίνδυνο να μην γνωρίζετε αν τελικά ναι ή όχι θα σα αποζημιωθούν ε, τα έξοδά σα ε, για κάποια, κάποιες στοιχείες περίθαλψη, εν πάση περιπτώσει. Εάν ζητάνε κάποια ασφάλεια, θα πρέπει να δεχτούν ένα σύστημα που να μπορέσει να παράσχει αυτή την ασφάλεια, γιατί αλλιώς θα επικρατήσει αυτό το στοιχείο της ε, ανασφάλειας. Εάν θέλετε ένα πιο ανοιχτό σύστημα πρέπει να δεχτείτε και την ε, ε, έλλειψη σιγουρία σχετικά με την αποζημίωση ή όχι. Αυτά σε σχέση με την πρώτη έγκριση δεν είναι μόνο ότι εμπλέκονται τα, τα κρατημέλη και αρμοδιότητε του, απλά οι ασθενείς τι θέλουν. θέλουν ασφάλεια σχετικά με την αποζημίωση, τότε το σύστημα θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει να γνωρίζουν αν θα γίνει η αποζημίωση. Μας λένε όλοι ότι θέλουμε σιγουριέ, λοιπόν πρέπει να έχουμε το αντίστοιχο σύστημα. Τώρα για την ευθύνη ναι, είναι ευθύνη του κράτους μέρους όπου γίνεται η ε, περίθαλψη, αλλά εγώ έχω και κάποιες απορίες. Ε, τα μεμονωμένα κράτη-μέλη σε ποιο βαθμό ε, θα μπορέσουν να δώσουν σαφείς και συγκρίσιμες πληροφορίες σε σχέση με άλλα 26 κράτη-μέλη. Απορώ εγώ αν γίνεται αυτό. Η συμβαστική AIDS προς τα αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει πάντως. Και από ό,τι κατάλαβα, από τον κατάλογο των αρμοδιοτήτων που ζητάμε από την Επιτροπή ε, αυτή είναι μία από τις ευθύνες, αυτό το άρθρο. Πάντως, ε, για να υπάρχει ασφάλεια και σε σχέση με... Ε, θα πρέπει η Επιτροπή Περιβάλλοντος να αναγνωρίσει την πραγματογνωμοσύνη μας στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστούμε. Ε, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μπραγκέτο, θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Γενικά να πω ότι υπήρξε πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες επιτροπές και υπάρχουν οι σωστές προϋποθέσεις ώστε να καταλήξουμε σε ευρεία συνένεση για τα εκρεμή ζητήματα, τα ζητήματα δική μας, δικής μας αρμοδιότητας. Ε, πολύ καλή συνεργασία είχαμε. Ε, εγώ ίδιος δεν συνηθίζω να υποβάλω τροπολογίες, ε, αλλά με τον Ούλε Κρίστανσον συντάξαμε από κοινού μια τροπολογία και την κυρία Λάμπερτ για την ε, πρώτερη έγκριση συγκεκριμένα. Έχει συζητηθεί επί μακρόν αυτό το θέμα της πρώτερης έγκρισης για το σύστημα υγειονομική περίθαλψης, όπως είπε και η κυρία Λάμπερτ, είναι θέμα ασφάλειας ε, ε, του ε, ασθενούς. Δηλαδή να ξέρει ότι μπορεί να πάει σε ένα άλλο κράτος μέλος, να λάβει την υγειονομική περίθαλψη και να επιστρέψει και να ξέρει ότι θα θα αποζημιωθούν οι δαπάνε του. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που έχουν άνεση οικονομική και μπορούν να το διακινδυνεύσουν. Άλλοι όμω δεν έχουν τόσο παχύ πορτοφόλι και θα πρέπει να ξέρουν ότι όντως θα πάρουν την έγκριση και όντως θα τους αποζημιωθούν, ε, αποζημιωθούν συγγνώμη, τα έξοδα για αυτή την υγειονομική περίθαλψη που τους παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον ασθενή. Και γι' αυτό ε, συμφωνώ για αυτή την τροπολογία, για την πρώτερη έγκριση. Αυτή η τροπολογία έχει κέρια σημασία μέσα στην οδηγία. Τέλος, επί της διαδικασίας. Ε, σχετικά με την ψηφοφορία. Για δύο λόγους άλλαξαν τα πράγματα. Πρώτον, γιατί ενημερώθηκα από τον πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας έστειλε επιστολή στην Επιτροπή Νομικών ε, Θεμάτων για το θέμα της νομικής βάσης. Δεν ανακοινώθηκε, δεν κοινοποιήθηκε η επιστολή, αλλά εγώ την έλαβα ε, και έλεγε ότι έχουν υποβληθεί διάφορες τροπολογίες στην Επιτροπή του που αποσκοπούν στην αλλαγή της νομικής βάσης με διάφορους τρόπους. Πρέπει να αποφανθεί η νομική επιτροπή λοιπόν για αυτά τα ζητήματα οπωσδήποτε. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο άλλος λόγος είναι ότι ε, δεν ήμουν εκεί στην προηγούμενη συζήτηση. Το έμαθα εγώ σήμερα ότι συζητήθηκε το θέμα των αρμοδιοτήτων μας σε σχέση με την αρμοδιότητα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας. Στο ενδιάμεσο διάστημα πρέπει να είμαι σε επαφή με τον κύριο Μπραγκέτο γιατί πρέπει να δούμε ακριβώς πώς επηρεάζει την κατάσταση στο θέμα της νομικής βάσης. Δηλαδή να ξέρουμε ποια είναι η άποψη της Επιτροπής μας για τις αρμοδιότητες μας για αυτό το θέμα σε σχέση με τις αρμοδιότητες ε, της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος. Τόσο χρήσιμο ήταν που κάναμε τη συζήτηση παρόλα αυτά ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό που υπάρχει ομοθυμία για αυτή την οδηγία. Αλλά αναβάλαμε την ε, ψηφοφορία και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το θέμα της νομικής βάσης και το θέμα της κατανομής των αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε επιτροπές. Αυτή την πρόταση κάνω εγώ. Κύριε Μπραγκέτο, θέλετε να συνοψίσετε τη συζήτηση. <clears throat> Εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω. Λοιπόν, θα πρέπει παρά τα σημαντικά αποτελέσματα που είχαμε να δούμε πώς θα επεξεργαστούμε καλύτερα τα άρθρα 72, 73, 74 θα τα κοιτάξουμε να τα βρούμε με ρία το ίδιο και για την τροπολογία για τις τροπολογίες 36 και 38 των πρασίνων τώρα για τα άλλα δύο ζητήματα οι θέσεις τη συναδέλφου για το πόσο μετριοπαθές είναι το άρθρο 8 Τέλος πάντων όμως εδώ πρόκειται για έναν συμβιβασμό, είναι το μάξιμουμ της συνένεσης που μπορέσαμε να πετύχουμε. Είναι αυτό το σημείο ισορροπίας που βρήκαμε. Για το 191 δεν υπάρχει καμία αντίρρηση ουσίας όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι για τον ασθενή να κατανοεί ότι ο γιατρός στον οποίο πηγαίνει ε, έχει μια εγγυημένη επαγγελματική κατάσταση. Το θέμα των επαγγελματιών όμως είναι το θέμα το οποίο εξετάζεται στην επόμενη οδηγία όπου προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα της εγγύησης, της επαγγελματικότητας, αυτού που παρέχει την υπηρεσία, αλλά δεν είναι η αναλυτική παρουσίαση εδώ του θέματος. Το συζητήσαμε και την άλλη φορά, το ζήτημα αυτό των αμοιβαίων ε, ε, ικανοτήτων, αν θέλετε τώρα αυτό να το, να το ξεκαθαρίσουμε και να το συζητήσουμε πριν από την αυριανή ψηφοφορία Μα τι να σας πω, αυτό είναι απόφαση και του πρόεδρου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μπραγκέτο. Ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Εγώ έκανα μία πρόταση να αφήσουμε χρόνο για να συζητήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και θα δούμε σύντο χρόνο τι θα γίνει. Απλά ο κύριο Μπραγκέτο μπορεί να μα πει συγκεκριμένα τι θα γίνει με την κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στι επιτροπέ στο ενδιάμεσο διάστημα να μα ενημερώσει. Δηλαδή περιμένοντα και την απάντηση για την νομική βάση. Τέλο πάντων προ το παρόν λίγη η συζήτηση. Πάμε τώρα στο... Επόμενο σημείο, δικό μου και αυτό, απαλλαγή 2007. Πολύ σύντομος θα είμαι. Μία τροπολογία έχω πάρει από την κυρία Στάουνερ. θέλει να προσθέσει το από κοινού με τα κράτη-μέλη και να συνεχίσει υλοποίηση ε, σχεδίου δράση για την περαιτέρω βελτίωση των συστημάτων ελέγχου και τη εποπτεία τη Ένωση. Θέλει να προσθέσουμε αυτό το κομματάκι, αυτή την αράδα από κοινού με τα κράτη-μέλη. Συμφωνώ, κυρία Στάνο, να το προσθέσουμε. Άλλε τροπολογίε δεν έχουμε. Θέλει κανεί το λόγο. Όχι είναι περίτη η συζήτηση, μπορώ να θεωρήσω. Ωραία. Πολύ απλά τα πράγματα. Προχωράμε με βήματα χ. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ταμείο Συνοχής, διατάξεις σχετικά με την δημοσιονομική διαχείριση. Κυρία Κρετή. Κύριε Κρετή, Γαμπριέλα. Report. The floor is yours. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλο αυτό το ζήτημα. Αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τη γραμματεία Θέλω έλεγα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην τροποποίηση αυτής της έκθεσης. Θέλετε να τα ξαναπώ όλα από την αρχή όμως αφού ήδη έχουν συμμετάσχει οι συνάδελφοι. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση αφού μου λέτε όχι, να ευχαριστήσω τη γραμματεία και σύμφωνα με το ότι αποφασίστηκε και την προηγούμενη φορά θα δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη για την απλούστευση των διαδικασιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τροπολογίες δεν υπάρχουν. Ε. Και ε, θα ψηφίσουμε αύριο. Λήξη και αυτή τη συζήτηση. Πάμε τώρα στο επόμενο σημείο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και του συντονιστέ σήμερα, άμα το ξέραμε ότι τόσο γρήγορα θα τα τελειώναμε όλα για την οδηγία για το χρόνο εργασία. Τέλο πάντων, η συμμεταχείριση αντρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελεία επαγγελματική δραστηριότητα. Ο κύριο Κοτσιλόβο, έχετε τον λόγο. Grazie Presidente, anch'io sarò molto breve, abbiamo già fatto la discussione generale. Λοιπόν, κάναμε εμεί αυτή τη συζήτηση για την ε, έκθεση γνωμοδότηση σε θεμελιώδης ε, αρχές είναι να έχουμε την, τον ορισμό μεταξύ συμβιόντων, συζύγων, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και αυτές οι αρχές σχετικά με τους ε, συντρόφους συμβίωσης κλπ. Ίσχυουν για όλες τις επιχειρήσεις για να έχουμε μία ισότιμη κάλυψη από κοινωνικής πλευράς. Και αυτό ισχύει για τον βασικό εργοδότη και όταν υπάρχει αρχή της υποχρέωσης τότε πέρα από τις ε, συζύγους και οι σύντροφοι συμβίωσης καλύπτονται. Εγώ θα έλεγα λοιπόν να δεχθούμε τις τρεις τροπολογίες της κυρίας Ρέντερ και την τροπολογία της κυρίας Μπάουερ που αναφέρονται στην οικογενειακή επιχείρηση και ενισχύουν τις ιδέες που ήδη εμπεριέχονται στην έκθεσή μου. Γνωρίζω ότι από την νομική υπηρεσία μας ζητείτε εάν συμφωνήσουμε σε αυτές τις τροπολογίες να κάνουμε μία γλωσσική επαλήθευση Χρωστάω μία απάντηση όμως στην κυρία Μπάουερ που είχε θέσει ένα ζήτημα ε, λέγοντας ότι σε πολλές ε, τροπολογίες εγώ έβαλα πολύ περιστόνισα πολύ περισσότερο τους συντρόφους συμβίωσης πέρα από τους, ε, τις και συμβοηθούντες συζύγους. Εγώ θα ήθελα σε όλα τα άρθρα ουσίας κάθε φορά που μιλάμε για συζύγους να μιλάμε για συζύγους και για τους συντρόφους συμβίωσης. Θεωρώ από νομικής πλευράς είναι σαφέστατο το πράγμα. Προτείνω λοιπόν το κείμενο έτσι όπως έχει παρουσιαστεί με την προσθήκη αυτών των τροπολογιών για την τελική αποδοχή του κειμένου. Ευχαριστώ πολύ. Αρχίζει η συζήτηση. Κανένας δεν θέλει το λόγο. Θα ψηφίσουμε αύριο λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Κοτσιλόβο. Α, έχουμε ακόμη ένα σημείο και το είχα ξεχάσει. Το θέμα της προφορικής ερώτησης για τα παιδιά των μεταναστών που έχουν μείνει στη χώρα προέλευσης. Θα θυμάστε ότι ως εισηγητής έχω οριστεί εγώ και αυτό γιατί είμαι πρόεδρος της Επιτροπής για τις προφορικές ερωτήσεις και τα ψηφίσματα ε, είναι η Επιτροπή που εκφράζεται είναι μέσω του Προέδρου. Η κυρία Μπλούμ αυτή η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία. Δεν θα ήθελα τώρα να κάνω παρουσίαση, διότι δεν έκανα εγώ τη δουλειά. Μιλάω εξ ονόματος της Επιτροπής και δίνω το λόγο στην κυρία Μπλούμ για να μας τα πει. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή και τον Στίβεν Χιούξ και τον Πίτερ για την βοήθεια που μας δώσανε. Εάν μου επιτρέπετε θα ήθελα να σας ε, πω τι στόχους είχα καταθέτοντας αυτή την ερώτηση. Η χώρα μου έχει πολλά προβλήματα με τα παιδιά που παραμένουν στη χώρα όταν οι γονείς μεταναστεύουν. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο είναι πάρα πολύ αρνητικό συνολικά στην κοινωνία. Τα τελευταία δύο χρόνια το φαινόμενο αυτό πήρε τεράστια έκταση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε στατιστικές σχετικά με την κατάσταση στα κράτη-μέλη για να δούμε πόσα παιδιά πλήττονται από αυτό το φαινόμενο, δηλαδή την αναχώρηση των γονιών τους που μετανάστευσαν για να εργαστούν σε μια άλλη χώρα. Στη Ρουμανία και αυτό με τη συμφωνίες συνεργασίας που έχουμε συνάψει με την κοινωνία των πολιτών κάναμε μία μελέτη και βάσει αυτής της μελέτης ε, διαπιστώσαμε ότι είναι περίπου 350.000 παιδιά τα οποία επηρεάζονται από αυτού του είδους ε, την ε, κατάσταση και ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των παιδιών έχουν μείνει εντελώς μοναχά τους, δεν υπάρχει κανείς μα κανείς να τα φροντίσει διότι έχουν μεταναστεύσει και οι δυο γονείς. Αφορά όλη την κοινωνία αυτό το φαινόμενο και τα παιδιά και τους γονείς φυσικά τα παιδιά είναι αυτά τα οποία πλήττονται άμεσα διότι δεν πάνε σχολείο, εγκαταλείπουν το σχολείο, υποφέρουν από κατάθλιψη και τα παιδιά αυτά των οποίων οι γονείς ε, έχουν οι πλησιέστεροι συγγενείς, έχουν φύγει, είναι εντελώς μόνα τους κλπ. Πολλές φορές προσπαθούν και να αυτοκτονήσουν. Έχουμε πολλές απόπειρες αυτοκτονίας παιδιών στην ε, Ρουμανία τα οποία είναι θύματα κοινωνικής και επίση από αυτή την κατάσταση δημιουργούνται και κοινωνικές ανισορροπίες. Πρέπει λοιπόν εμείς να φανταστούμε συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά και αυτές τις οικογένειες ούτω ώστε να εγγυηθούμε το μέλλον της, των μελλοντικών ευρωπαϊκών γενεών. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ε, είμαστε, έχουμε περάσει στην πολυγλωσία γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Λάμπερτ επίσης έχει τον λόγο. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο που έθιξε το ζήτημα. Εγώ έχω, η ομάδα μου έχει μία σειρά τροπολογίες που δεν αλλάζουν την ουσία αλλά το ύφο. και ξεκαθαρίζουν βέβαια στο πεδίο εφαρμογή για να ξεκαθαρίσουμε πως μιλάμε για παιδιά υπηκόους της Ένωσης και όχι ανά τον κόσμο γιατί είναι άλλη αυτή η υπόθεση πολύ μεγαλύτερη και επίσης για να ξεκαθαρίσουμε πως πρόκειται για έναν κίνδυνο και δεν είναι αυτόματο αυτό για όλα τα παιδιά. Είναι ένας κίνδυνος που διατρέχουν κάποια παιδιά. Αυτή είναι η βάση των αλλαγών που προτείνουμε. Δεν αλλάζει πολύ ουσία. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό να εξετάσουμε το πλαίσιο της μελέτης, οπότε ελπίζω να λάβουμε θετική απάντηση στο ερώτημα. Σας ευχαριστώ η κυρία Τομασέφσκα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις ερωτήσεις αυτές και για το ότι ζητάμε απάντηση από την Κομισιόν. Το πρόβλημα των παιδιών χωρίς γονείς στην Πολωνία είναι πολύ σοβαρό, ίσως να υπάρχει και σε άλλες ε, χώρες και πρέπει να λυθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα κλείσει λοιπόν αυτή η συζήτηση. Βεβαίω πρόκειται για πρωτοβουλία της Επιτροπής μας. Ε, συμφωνώ, είναι πολύ σημαντική και οι τρεις ομιλήτριες το τόνισαν αυτό. Πρέπει πράγματι το ζήτημα αυτό να κατατεθεί και να αναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία. Λοιπόν, λίγες τροπολογίες έχουν κατατεθεί αργά σήμερα και ελπίζω να καταφέρουμε να συμφωνήσουμε πριν την ψηφοφορία αύριο. Ελπίζω να συμφωνήσουν σε αυτές τις τροπολογίες πολιτικές ομάδες για να έχουμε ένα σαφές μήνυμα δήλωση αν θέλετε της Επιτροπής μας όταν θα πάμε στην επόμενη Ολομέλεια θα ήταν καλό κάτι τέτοιο τελειώσαμε λοιπόν με αυτό το θέμα με την προφορική ερώτηση και τα ψήφισμα οπότε νομίζω ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής ημερήσιας διάταξης σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας για το ενδιαφέρον που δείξατε συνεδριάζουμε πάλι αύριο αύριο ψηφοφορία παρακαλώ φέρτε τις κάρτες σας και ευχαριστώ και τους διερμηνείς. δεν θα γίνει η συνεδρίαση των συντονιστών. Μπορούσαμε να την κάνουμε από ό,τι φαίνεται, αλλά δεν το ξέραμε, οπότε λύεται η συνεδρίαση. Γεια σας.